Hello everyone. Καλημέρα σε όλους και όλες. Θέλουμε να παραμείνουμε στο χρονικό μας πλαίσιο. Καθίστε παρακαλώ. Και θυμαστείτε να ακούσετε τις πολυδιαφέρουσες παρεμβάσεις και να είστε έτοιμοι να θέσετε ερωτήσεις. Καλώς ήλθατε όλοι και όλες στην ακρόασή μας για την ε, παροχή ασύλου. Το θέμα της πρόσβασης σε αποτελεσματική προσφυγή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αυτό θα είναι το πρώτο θέμα που θα μας απασχολήσει στο πρώτο αυτό απογευματινό πάνελ. Το δικαίωμα για πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή προβλέπεται στο κεφάλαιο θεμελιωδών δικαιωμάτων της Χάρτας που έχει ενσωματωθεί στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι αυτό είναι κομμάτι της Συνθήκης. Και να σας αναφέρω δύο λόγια για τη σημασία του δικαιώματος αποτελεσματικής προσφυγής. Θεωρείται ότι είναι μία από τις βασικές αρχές δικαίου, περιλαμβάνεται στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος αυτού του δικαιώματος είναι να εξασφαλιστεί η ουσία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σε οποιαδήποτε μορφή και αν καθαγιάζονται στο εθνικό δίκαιο. Υπάρχει η πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου, του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε σχέση με την πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή που αναφέρει ουσιαστικά η νομολογία αυτή. Λέει ότι μία προσφυγή είναι αποτελεσματική αν επιτρέπει την ε, εφαρμογή κάποιου δικαιώματος ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, τουλάχιστον δίδει μία αποτελεσματική θεραπεία για το δικαίωμα αυτό. Θα συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα με τους καλεσμένους μας. Ξεκινώ καταρχήν κυρία Σαμπίνα Χεξκίλ που είναι από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Ακολουθεί ο κύριος ε, Σέρζ Μποντάρ, πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Αντιδικιών Αλλοδαπών, μέλος του Συμβουλίου Επικρατείας, λέκτορας στο Ίδρυμα Ευρωπαϊκών Σπουδών και Συνομική Σχολή του Πανεπιστημίου ULB, Βέλγιο. Μετά ο κύριος Νίλ ε, Φέιλζον, διευθυντής του ΕΜΚΟ Αντίτους, προσκεκλημένος λεκτόρας του Πανεπιστημίου της Μάλτας και υπεύθυνος του μπλοκ παρακολουθήσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα συλλου, ΕΑΣΟ, και ο κύριος ε, τέλος ο Δόκτωρ Μάρτεν Ντεν Χέιρ, μέλος της Επιτροπής Μέιερς, μόνιμη Επιτροπή Εμπειρογνωμών και το Διεθνές Δίκαιο σε θέματα μετανάστευσης, προσφύγων και ποινικού δικαίου. Κυρία Χέξκιν, για την κατάσταση της νομολογίας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση της αποτελεσματικής πρόσβαση, αποτελεσματική πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα ξεκινήσει. Παρακαλώ. Το, κυρία Πρόεδρε. Η πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή διασφαλίζεται από το άρθρο 47 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και αυτό ε, σε ε, οποιονδήποτε χέρι των δικαιωμάτων ε, που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί μέρος του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ισχύει σε τη ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας του Δεκέμβριο του 2009. Όμως υφίστατο ήδη, προϋπήρχε δηλαδή βάση νομολογίας ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που είναι ε, σταθερή εδώ και 25 έτη. Είναι η αρχή λοιπόν της αποτελεσματικής προσφυγής που αποτελεί ε, ε, ευρεία αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που απορρέει από την ομολογία ε, των, ευρωπαϊκών, των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και ρητά αναφέρεται στα άρθρα 6 και 13 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αυτή η αρχή εφαρμόζεται επί όλων των δικαιωμάτων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών. Η υπόθεση Jones 1986, ε, ε, όπου για πρώτη φορά αναφέρεται ρητά, το δικαίωμα το οποίο απορρέει από την ε, η ευρωπαϊκή υπηκότητα, ε, την εσωτερική αγορά, καθώς επίσης ε, και την ελεύθερη εκκίνηση μέσα στον χώρο δικαιοσύνης και ελευθερίας, κυρίως σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά το άσυλο και εδώ βεβαίως ε, υλοποιείται ε, και ε, εφαρμόζεται το δίκαιο από τα χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως στις νομολογίες των κρατών μελών θα πρέπει να βρούμε την πραγματική δυνατότητα σε αποτελεσματική προσφυγή και αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τα εθνικά δικαϊκά συστήματα. Όντως, ελήψη νομοθεσίας του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ενωσιακό επίπεδο, το κάθε κράτος μέλος θα είναι αυτό που θα καταδείξει την αρμόδια αρχή, καθώς επίσης και τις ε, ε, προβλεπόμενες ε, διαδικασίες πρόσβασης, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται στους ενδιαφερόμενους τα δικαιώματα, έτσι όπως αυτά απορρέουν τη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το ε, και από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οποτεδήποτε ε, έχουμε παραβίαση αυτής της τελευταίας μορφής δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, συμμετέχει στην διαδικασία απονομής ε, δικαίου όσον αφορά το άσυλο. Δηλαδή συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές στα πλαίσια της ε, προδικαστικής διαδικασίας απαντώντας σε προδικαστικά ερωτήματα όσον αφορά την ερμηνεία νομοθεσίας ευρωπαϊκής καθώς επίσης και όσον αφορά το παράγωγο δίκαιο και βεβαίως μπορεί κατά αυτήν την έννοια να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, και ευρωδικαστικό ερώτημα το οποίο αναφέρεται ε, το πραγματικό δίκαιο. Για παράδειγμα, μπορώ να σας πω για τον τομέα που μας ενδιαφέρει. Μπορούμε λοιπόν να αναφερθούμε ε, σε, στην απόφαση Σάμπα Τιούρφη 28 Ιουλίου του 2011 ε, που αφορά την οδηγία 205-85 όσον αφορά τα ε, ελάχιστα στάνταρ για την δυνατότητα προσφυγής στο καθεστώς πρόσφυγα στο κράτος μέλος. Ο κύριος Σαμαντιούφ είναι πίκος της ε, Μαυριτανίας ε, και η εισήγαγε έτοιμα για διεθνή προστασία στο Λουξεμβούργο στη διάρκεια της συνέντευξής του δήλωσε ότι εγκατέλειψε την χώρα του, την Μαυριτανία, έτσι ώστε να ξεφύγει από ένα καθεστώς σκλαβιάς και ότι επιθυμεί να εγκαταθεστεί στην Ευρώπη για να ζήσει με καλύτερες συνθήκες και να μπορέσει να ε, ιδρύσει οικογένεια είπε ότι για να μπορέσει να φύγει από την Μαυριτανία έκλεψε 3.000 ευρώ από το αφεντικό του ε, και φοβάται ότι εάν επιστρέψει στην Μαυριτανία, στην θα τον κυνηγήσει και θα τον σκοτώσει το αφεντικό του. Ε, δύο πράγματα έκανε το ε, Λουξεμβούργικο Δικαστήριο. Πρώτον, αποφάσισε να εξετάσει το αίτημα του κυρίου ε, αυτού ε, σε γρήγορη διαδικασία, επιτυχημένη διαδικασία. Στα πλαίσια όμως της διαδικασίας αυτής απέρριψε το θέμα επί της ουσίας λέγοντας ότι ο κύριος Σαμπαντιούφ ε, είχε υποβάλει πλαστό διαβατήριο και ότι οι λόγοι τους οποίους είχε αναφέρει στα πλαίσια του αιτήματό του αφορούσαν οικονομικά αίτια και επομένως δεν μπορούσε να του δοθεί η προστασία που ζητούσε. Ο κύριος Σάμπαντιούφ ε, προσέφυγε κατά της ε, απόφασης αυτής. Το, ε, Λουξεμβούργιο, το Λουξεμβουργικό δίκαιο προβλέπει ότι όταν έχει ολοκληρωθεί στα πλαίσια επιταχυμένης διαδικασίας η μελέτη ενός αιτήματο προστασίας ότι λέει είναι ε, δυνατή η προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο αλλά η προθεσμία, ε, η προθεσμία υποβολής ε, είναι πιο σύντομη από ότι εάν δεν είχε ακολουθηθεί η επιταχυμένη αλλά η απλή διαδικασία. Επίσης, το δίκαιο του Λουξεμβούργου αποκλείει την δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης για επιταχυμένη διαδικασία μελέτης του αιτήματος. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην περίπτωση Σαμπαντιούφ, ε, ε, συγγνώμη, το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου είχε αμφιβολίες όσον αφορά το αίτημα του κυρίου Σαμπαντιούφ. Ε, δηλαδή είχε δικαίωμα να κάνει την προσφυγή και επίσης στα πλαίσια της προσφυγής αυτής το αίτημα το οποίο αιτείται είναι συμβατό με την δυνατότητα αποτελεσματικής προσφυγής και απευθύνεται σχετικά ερωτήματα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρώτον, όσον αφορά ε, την οδηγία, εκεί ρητά αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική προσφυγή κατά της απόφασης που αφορά το αίτημα ε, ασύλου. Η ερώτηση λοιπόν ήταν η απόφαση ε, να συζητηθεί το θέμα αυτό με επιταχυμένη διαδικασία ήταν αποδεκτό. Βεβαίως όταν βλέπει κανείς τη διατύπωση ε, φαίνεται σαφές ε, ότι η απόφαση είναι εφικτή, δηλαδή η απόφαση για επιταχυμένη διαδικασία. Όμως, κατά την ερμηνεία του δικαστηρίου, διορθώνει η ομιλήτρια, αλλά ε, στην ουσία αυτή η απόφαση για επιταχυμένη διαδικασία προετοιμάζει, προλιένει το έδαφος για την τελική απόφαση, για το κατά πόσο δηλαδή ή ε, το αίτημα ε, για την, για, αυτή, αυτή, αυτή, το, για αυτό καθε αυτό το καθεστώς ασύλου θα γίνει δεκτό ή όχι. Επομένως, αυτή η προπαρασκευαστική διαδικασία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο χωριστής προσφυγής. Επομένως ε, δεν υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά την οδηγία. Δεύτερο ερώτημα, ε, όλη αυτή η διαδικασία είναι συμβατή με το δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή. Κατά αυτήν την έννοια το ε, δικαστήριο βασίστηκε σε υφιστάμενη νομολογία που λέει ότι δεν είναι απαραίτητο για να υπάρχει αποτελεσματική προσφυγή όλες οι αποφάσεις οι προπαρασκευαστικές να μπορούν να εφεσιβληθούν αρκεί να ε, μπορεί να εφεσιβληθεί η τελική απόφαση. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό ε, την προκειμένη περίπτωση είναι ο λόγος για τον οποίο απορρίπτεται ε, το αίτημα προστασίας. Αυτή η απόφαση θα πρέπει ενδελεχώς και σε βάθος να μελετηθεί από τον ε, δικαστή. Σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου, ε, το αιτιολογικό για την επιλογή της επιταχυμένη διαδικασία στην ουσία ε, είναι περίπου ταυτόσιμο με το σκεπτικό της απόρριψης του ιδίου του αιτήματο. Ε, αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή ε, τα πλαστά διαβατήρια του κυρίου Σαμπαντιούφ, τους λόγους που επικαλέστηκε κτλ. Όλα τα στοιχεία αυτά συζητήθηκαν από το δικαστήριο και από τους δικαστές στα πλαίσια της διαδικασίας αποτελεσματικής προσφυγής. Και επομένως, ε, καταλήγουμε ότι δεν είναι αποδεκτό βάση ε, της αρχής την πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή εάν ε, το δίκαιο του Λουξεμβούργου ερμηνευθεί με τρόπον ώστε να μην μπορεί να εφεσιβληθεί η απόφαση για επιταχυμένη διαδικασία διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούσε να γίνει η ενδελεχής προβλεπόμενη μελέτη ε, του θέματος αυτού στα πλαίσια της ε, ε, τελικής συζήτησης για την αποτελεσματική προσφυγή. Επομένως, μπορούν να μπορεί να ελεχθεί η απόφαση αυτή. Και επομένως η απόφαση ε, για επιλογή της επιταχυμένης ε, διαδικασίας μπορεί να μην αποτελέσει αντικείμενο χωριστής προσφυγής. Επίσης, το δικαστήριο αναφέρθηκε στα άλλα δύο διαδικαστικά ζητήματα. Πρώτον, το πρόβλημα της προθεσμίας ε, υποβολής ε, προσφυγής ε, που είναι 15 ημέρες μονάχα για την επιταχυμένη διαδικασία και εκεί απεφάνθη ότι εξαρτάται από τις συνθήκες. Δηλαδή, ε, μία τέτοια προθεσμία ε, είναι, θεωρείται ε, λογική, θα πρέπει αυτή να ελεγχθεί από τον εθικό δικαστή, ο οποίος θα αποφανθεί εάν το περιθώριο των 15 ημερών δίνει όλες τις δυνατότητες των προσφεύγοντα. Διαπιστώνει πάντως το δικαστήριο κατά την έννοια αυτή ότι ε, τα, ε, τα κράτη-μέλη αλλά ε, και οι ετούντες άσυλο έχουν κάθε συμφέρον να ληφθούν γρήγορα οι τελεσίδικες αποφάσεις και επομένως είναι μάλλον ευνοϊκό το δικαστήριο απέναντι σε μια γρήγορη διαδικασία λήψης απόφασης. Επίσης, το δικαστήριο απεφάνθη ότι υπάρχει, ε, ε, ε, ότι το γεγονός ότι υπάρχει μόνο μία δυνατότητα προσφυγής είναι λογική, δηλαδή μπορεί να γίνει προσφυγή σε ένα δικαστήριο μονάχα. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να κρατήσω λίγο χρόνο για τη συζήτηση και ενδεχομένως ερωτήσεις και μπορείτε να απαντήσετε ενδεχομένως απαντούσα στις ερωτήσεις να προσθέσετε και κάτι ακόμα αν θέλετε, αλλά τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σέρζ Μπονταρ, ο οποίος θα μιλήσει για τις αποκλίνουσες ερμηνείες ε, στα κράτη-μέλη που σημαίνουν διαφορετική πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή. Merci, Madame la Présidente. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω την παρέμβασή μου δίνοντας σας μια πρακτική αν θέλετε διευκρίνηση αντίθετα από τους περισσότερους ε, ομιλητές σήμερα εγώ δεν εκπροσωπώ κανένα θεσμό, κανένα οργανισμό ε, αυτό ίσως να είναι και πλεονέκτημα σας μιλώ βάσει της δικής μου προσωπικής εμπειρίας ως Προέδρου για πολλά χρόνια ενός ε, δικαστηρίου κατά κάποιο τρόπο το οποίο είχε σαν στόχο να εξασφαλίσει την ε, αποτελεσματική προσφυγή σε αλλοδαπούς. Και εδώ θέλω να σταθώ σε μια προβληματική που αντιμετώπισα για πολύ καιρό μέσα στην ίδια μου τη χώρα και αυτή η προβληματική αφορά την ανάγκη να ενσωματώσουμε τα αποτελέσματα της πρόσβασης στην αποτελεσματική προσφυγή σε μια διαδικασία εναρμόνισης <clears throat> και ιδίως όταν αυτή η διαδικασία εναρμόνισης γίνεται προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος σε ό,τι αφορά την παροχή ασύλου. Όταν μιλάμε λοιπόν για εναρμόνιση για τα θέματα του ασύλου, σε τι αναφερόμαστε. Είναι απλή ιδέα ότι κάποιος ο οποίος ζητά το άσυλο θα πρέπει να έχει ισοδύναμες πιθανότητες επιτυχίας ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία εισάγει την αίτησή του. Και όταν μιλάμε για αποτελεσματική προσφυγή, και εκεί η βασική ιδέα είναι πολύ απλή, η αρχή αυτή προκύπτει από το άρθρο 47 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, δηλαδή ότι οποιαδήποτε ατομική απόφαση η οποία απορρίπτει μία αίτηση ασύλου θα πρέπει να υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον ανεξαρτήτου δικαστηρίου. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν τόσα ανεξάρτητα δικαστήρια τουλάχιστον όσο και χώρες μέλη και στην πραγματικότητα περισσότερα γιατί σε πολλές χώρες η αρμοδιότητα για τα θέματα ασύλου έχει διαβιβαστεί σε ε, αποκεντρωμένα δικαστήρια, δικαστήρια με πολλά τμήματα. Στην περίπτωση του Βελγίου υπάρχει μονάχα μία δικαστική περιφέρεια, αλλά υπάρχουν πολλά μονοεδρικά τμήματα τα οποία εκδικάζουν τέτοιες υποθέσεις και έχουμε στην πραγματικότητα 30 διαφορετικούς δικαστές οι οποίοι αποφασίζουν για τα θέματα αυτά, κάτι το οποίο μπορεί να δώσει λαβή σε 30 διαφορετικές νομολογίε. Τώρα, δεν είναι πολύ εύκολο να πείτε σε κάποιον να αποφύγετε τον τάδε τον β δικαστή. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν είναι πολύ σημαντικά για τα θέματα του ασύλου η ανάγκη εναρμόνισης υπάρχει για πάρα πολλά νομικά θέματα, αλλά στο θέμα του ασύλου είναι σημαντική η εναρμόνιση λόγω του ιδιαίτερου βάρους που υπάρχει στην περίπτωση αυτή στην διακριτική ευχαίρεια ερμηνείας. Όταν μιλάμε για ερμηνεία μιλάμε για υποκειμενικότητα. Αυτή η υποκειμενικότητα εμφανίζεται καταρχήν στον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζονται τα πραγματικά στοιχεία. Πολύ σπάνια κάποιο έρχεται με αποδείξεις ότι καταδιώκεται. Εγώ από την πείρα μου μπορώ να σας πω ότι γενικά κάποιος ο οποίος έρχεται με την απόδειξη ότι τον καταδιώκουν στη χώρα του, αυτό φαίνεται κάπως σάπιο, δηλαδή κάτι κάπως φαίνεται αυτό. Αυτό είναι η πρώτη αντίδραση που θα είχε ο υπεύθυνο προστασία όταν αντιμετωπίζει κάποιον ο οποίο φέρει μαζί του τις αποδείξεις. Επομένως συνήθω είναι ελάχιστα τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει ένα ετών άσυλο όταν υπάρχουν είναι πολύ δύσκολο να ξέρει κανείς ότι είναι αυθεντικά και γνήσια και γενικά δεν έχει πραγματικά τη δυνατότητα να ελέγξει και να επαληθεύσει απόλυτα την ακρίβεια αυτών των στοιχείων. Τι κάνουμε λοιπόν. Κάνουμε το λεγόμενο, τη λεγόμενη εξέταση αξιοπιστίας. Και εδώ εμπλέκεται πάρα πολύ η υποκειμενικότητα. Τον πιστεύω, δεν τον πιστεύω. Πάρα πολλές αιτήσει απορρίπτονται επί τη βάση αυτή. Μπορεί να σας φαίνεται μια λογική αρχή, αλλά η δική μου εμπειρία επί 20 χρόνια, οι περισσότερες αποφάσεις απόρριψης μιας αίτησης ασύλου είναι γιατί δεν μας αρέσει η φάση ενός ανθρώπου, δεν τον θεωρούμε αξιόπιστο. Και επιπλέον στα θέματα ασύλου η υποκειμενικότητα υπησέρχεται στην αναγνώριση ορισμένων βασικών στοιχείων. Γιατί και εκεί τα πράγματα είναι υποκειμενικά. Βάση της συμβάσης της Γενέβης ένας πρόσφυγας είναι κάποιος ο οποίος έχει λόγο να πιστεύει, ένας που ζητάει άσυλο, είναι κάποιος που έχει λόγο να πιστεύει ότι καταδιώκεται. Αλλά και αυτό είναι κάτι το, το αντικειμενικό. Το να πούμε ότι ένας φόβος είναι λογικός ή όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο το κρίνει αυτός ο οποίος πρέπει να πάρει μια απόφαση υπάρχει και στην ίδια την έννοια μια εγγενής πηγή υποκειμενικότητας. Η πρόκληση λοιπόν της αποτελεσματικής προσφυγής μέσα στο πλαίσιο αυτό και θα σας μιλήσω για τα θέματα ερμηνείας των νομικών ενιών. Στην πράξη η κύρια πρόκληση για τα θέματα αυτά που εμπλέκουν μεγάλη υποκειμενικότητα η, η πραγματική πρόκληση είναι να μπορέσει αυτός που ζητεί το άσυλο να δώσει συνεκτικά μηνύματα σε αυτόν ο οποίος θα λάβει την απόφαση. Και δεν είναι προφανές αυτό ότι μπορεί να το κάνει μέσα στην χώρα στην οποία ζητά το άσυλο. Επίσης πρέπει να υπάρξουν συνεκτικά μηνύματα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει κάποια δυνατότητα εναρμόνισης και επίσης μηνύματα συνεκτικά σε σχέση με την εναρμόνιση των πρακτικών που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από το Ευρωπαϊκό Διδακτικό Πρόγραμμα για τα θέματα αυτά ή μέσα από τις, από τους, τις ενώσεις των δικηγορικών συλλόγων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αν δεν θέλουμε να υποσκάψουμε όλη αυτή την προσπάθεια της εναρμόνισης. Η, τα δικαστήρια προσφυγής, τα δικαστήρια τα οποία είναι αρμόδια για τις προσφυγές, προσφυγές, να μην δίνουν αντιφατικά μηνύματα από τη μία χώρα στην άλλη. Πώ θα το πετύχουμε αυτό. Δεν υπάρχει κάποια πανάκια στα θέματα αυτά, αλλά πιστεύω ότι βάσει εμπειρία μου υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνε οι οποίοι μπορούν να μα βοηθήσουν σε αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνω μια σαφή διαφοροποίηση μεταξύ του ρόλου του δικαστή και των διοικητικών αρχών. Πρέπει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε ένα, όπως λέγω, κύκλωμα πλήρους ποιότητος από τον διοικητικό υπάλληλο μέχρι το δικαστή και δεν υπάρχει περίπτωση να κληθεί ο δικαστής να κάνει και πάλι την ίδια δουλειά που κάνει ο διοικητικό υπάλληλο. Αυτή είναι μια πρώτη ιδέα. Μια δεύτερη ιδέα είναι το να δώσουμε επίσημο και τυπικό χαρακτήρα στις διαδικασίες πρωτοβάθμιας εξέτασης. Γιατί αυτή η τυποποίηση είναι και μια απαράγραπτη προϋπόθεση για να βγούμε από αυτό που θα λέγαμε η τυραννία της υποκειμενικότητας. Δεν είναι λοιπόν θέμα απλώς καλής θέλησης, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες ρήτρε ε, σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο εκτιμά κανείς τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία μιας αίτηση ασύλου και μπορεί να αιτιολογήσει μια απόφαση. Και αυτή η... ο τυπικός χαρακτήρας είναι επί πάρα πολύ σημαντικός για να μπορέσουμε να περάσουμε σε ένα δεύτερο επίπεδο, να έχουμε ένα πιο τυπικό χαρακτήρα στον τρόπο με τον οποίο ασχεί το δικαστικό έλεγχο της αποφάσης παροχής ασύλου ο αρμόδιος δικαστής. Είναι ένα απλό ερώτημα πώς αυτά τα οποία σήμερα λειτουργούν σε πρακτικό επίπεδο, πώς θα πρέπει να μεταφραστούν σε νομικές διατάξεις. Και θα κλείσω με ένα κάπως εικονοκλαστικό ερώτημα, ιδίω ω πρώην πρόεδρο διοικητικού δικαστηρίου. Το ερώτημα είναι ποιο ελέγχει τους ελέγχοντε. Ο δικαστή ελέγχει τι διοικητικέ αρχές. Ποιο ελέγχει το δικαστή. Στι περισσότερε χώρες είναι σαφέ. Αυτό ο οποίο ελέγχει το δικαστή είναι ένα ανώτερο δικαστήριο. Υπάρχει αυτή η πυραμίδα των δικαστηρίων που είναι από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο και φτάνει μέχρι τον Άριο Πάγο. Αλλά δεν είμαι πεπισμένος ότι στα θέματα ασύλου αυτή η η ιεραρχία των δικαστηρίων είναι πλήρως οργανωμένη σε όλα, τα, σε όλα τα κράτη και αυτό το οποίο γνωρίζω πολύ καλά είναι ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή η πυραμίδα γέρνει. Είναι διαφορετικού χαρακτήρα σε κάθε χώρα δεν υπάρχει κορύφωση στις πυραμίδες αυτές. Κάθε χώρα έχει μια διαφορετική μορφή. Ένα προδικαστικό ερώτημα το οποίο μπορεί να τεθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να είναι ένας τρόπος για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια ενοποίηση και εναρμόνιση. Δεν μπορούμε όμως να θεωρήσουμε ότι αποτελεί αυτή η προδικαστική ερώτηση ερώτημα, ε, τρόπο ελέγχου της ε, απόδοσης δικαιοσύνης από τα υποκείμενα δικαστήρια. Μπορεί να φανταστεί τώρα κανεί να υπάρχουν εσωτερικοί έλεγχοι ποιότητα των δικαστηρίων, όπως γίνεται στις εθνικές διοικήσει. Αφήνω ανοιχτό αυτό το ερώτημα, γιατί εδώ προσκρούμε και στο θέμα της ανεξαρτησίας των ε, δικαστικών, που είναι ένα πρόβλημα μεγάλων διαστάσεων που δυσκολεύει και την ποιότητα εκδίκασης από τα δικαστήρια. Ευχαριστώ και μένω εδώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much. And now... Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ακούσουμε τον δόκτωρα Νίλ Φάλζον, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν για την πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή στις ε, διάφορες οδηγίες και στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλησπέρα σας. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών που μου ζήτησε να μιλήσω σε αυτή την τόσο σημαντική ακρόαση. Μια ακρόαση η οποία έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Από την πείρα μα, ε, ω μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούμαστε με θέματα ασύλου και ε, προσφύγων, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική ε, η, στο, η, αυτό το κοινό σύστημα σύλλου ε, αλλά ταυτόχρονα και επικίνδυνη, διότι ε, μπορεί ε, να αξιολογούμε το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλειστικά μόνο για λόγους ασφαλείας, διαχείρισης συνόρων και όλο και πιο αρνητικής αίσθησης του κοινού. Είναι πολύ δύσκολο να αναλύσουμε το δικαίωμα πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή και τον τρόπο με τον οποίο μεταφράζεται στα διάφορα νομικά μέσα και στις δικαστικές αποφάσεις, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από τις τεχνικές διαπραγματεύσεις και να καταλάβουμε τι επιπτώσεις έχουν οι οδηγίες για τους ετούντες άσολο, για τους πρόσφυγες και για τους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί τους αλλά δουλεύουν και για αυτούς. Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα λοιπόν. Πού είναι σημαντική η πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή και ποιες είναι οι καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για την πρόσβαση σε αυτά τα μέσα. Σε ένα διεθνέ πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή έχει καθοριστεί ω κάτι το οποίο έχει στόχο να εφαρμόζει την ουσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών με οποιαδήποτε μορφή και αν εμφανίζονται, ώστε να διασφαλίζονται στην εσωτερική δημόσια τάξη. Υπάρχουν αρκετέ ε, αποφάσεις από διεθνή και περιφερειακά δικαστήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, τις οποίε γνωρίζουμε. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η προσφυγή να είναι εύκολη, αποτελεσματική στην πράξη, προσβάσιμη, αμερόληπτη, ανεξάρτητη, να μπορεί να εφαρμόζεται και να πρέπει να οδηγεί σε πάυση ή σε ε, διόρθωση για παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δικαίωμα στην αποτελεσματική προσφυγή είναι εγγεγραμμένο στο άρθρο 47 της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το δικαστήριο πολύ συχνά λέει ότι είναι μια βασική αρχή του κοινοτικού δικαίου που απορρέει από τις ε, ε, συνταγματικές παραδόσεις που είναι κοινέ στα κράτη-μέλη και έχει εγγραφεί στα άρθρα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. η προφανής πρόσβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα ενισχύσει και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτών. Αλλά να δώσουμε μια ουσία στην πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή και να την ε, ε, θέσουμε στις διάφορες εκτυχίε, οι οποίες μας ενδιαφέρουν στη σημερινή ακρόαση. Αν δούμε τα διάφορα μέσα ασύλου που έχουμε, θα δούμε ότι ο βασικός όρος του δικαιώματος σε αποτελεσματική προσφυγή χρησιμοποιείται κυρίως στα πλαίσια της διαδικασίας ασύλου. Το κεφάλαιο 5 της ε, διαδικασίας, το εισοδηγία για τις διαδικασίες, μας δίνει διάφορες αποφάσεις από τα κράτη-μέλη και το πώς υποχρεούνται να εφαρμόσουν το δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή. Περιλαμβάνονται και αποφάσεις ε, ε, για τα σύνορα και αποφάσεις οι οποίες ε, μας οδηγούν στο να μην εξετάσουμε περαιτέρω κάποια θέματα. Όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή έχουμε διαπραγματεύσεις για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τροποποιήσουμε την οδηγία αυτή, αλλά δεν θα σταθώ σε αυτές αυτή τη στιγμή. Παρά το γεγονός ότι στην οδηγία αυτή ε, βρίσκουμε συγκεκριμένη διατύπωση πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή, υπάρχουν πολλές άλλες περιπτώσεις όπου ε, η πρόσβαση αυτή που είναι τόσο σημαντική για τους ετούντες έσυλο ε, μπορεί να εμφανίζεται. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι ετούντε άσυλο αντιμετωπίζουν αποφάσεις που λαμβάνονται από κυβερνητικές αρχές και που επηρεάζουν μία ή περισσότερες πτυχές τη ζωή του. Το να επισημάνουμε αυτές τις πτυχές ε, μας ενδιαφέρει επειδή θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αποφάσεις σε ένα πλαίσιο το οποίο ε, είναι αντίστοιχο των αποτελεσματικών κριτηρίων προσφυγής. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις οι οποίες ε, είτε ατομικά είτε συλλογικά απαγορεύουν σε τούντες άσυλο να διασχίσουν τα εξωτερικά σύνορα εκτός και αν διαθέτουν ε, ταξιδιωτικά έγγραφα. Ε, μας οδηγούν στο να κάνουμε ε, αποτελεσματικό έλεγχο για να δούμε κατά πόσον συνάδουν με το δικαίωμα στην αίτηση ασύλου και προστατεύονται από τη χάρτη των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν επίσης κάποια μέτρα τα οποία υιοθετούνται στην ανοιχτή θάλασσα από τα κράτη-μέλη ε, ατομικά στα πλαίσια των κοινών περιπελειών και επιχειρήσεων. Σαφώς εδώ ε, η Frontex ε, και κάποιες ε, ανησυχίες που αναφέρονται από τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας έρχονται κατά νου. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να μιλάμε για πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή οι αιτούντες έσυλο καλύπτονται τεχνικά από την οδηγία για την υποδοχή προσφύγων. Η πρόσβαση σε αποτελεσματικά μέτρα επίσης είναι πολύ σημαντική για αυτό το τομέα. Η οδηγία δίνει ε, αρκετή διακριτική ε, ευχέρεια στα κράτη-μέλη και μπορεί τα κράτη-μέλη να αποφασίσουν να μειώσουν ή να αποσύρουν ε, τις διάφορες συνθήκες υποδοχής. Στο κεφάλαιο 5 υπάρχει και το δικαίωμα άσκηση άφεση από πλευρά των ετούντων άσυλο, αλλά υπάρχουν πολλά πρακτικά θέματα που μα αποσχολούν. Τι πληροφορίε δίνονται καταρχά στου ετήνοντε άσυλο για την επέκταση των δικαιωμάτων του βάτη τη οδηγία. Ε, είναι ενήμεροι ότι μπορούν να κάνουν προσφυγή. Η έφεση για μια τέτοια απόφαση ε, έχουν δοθεί γραπτό οι πληροφορίε ή με ποιο άλλο τρόπο. Τι γλώσσα χρησιμοποιήθηκε για να δοθούν οι πληροφορίε. Η συνήθις έκφραση που έχουμε στις οδηγίες ε, στη γλώσσα την οποία υποτίθεται ότι κατανοούν οι αιτούντες άσολοι είναι σχεδόν ανόητη. Και ορισμένε φορές είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι δικαιώματα έχουν και το γεγονό ότι η δυνατότητά του για έφεση θα πρέπει να του δίνεται γραπτός και σε διάφορες γλώσσες. Τα θέματα αυτά αποκλείουν αποτελεσματικά και αγραμμάτους ανθρώπους ή ανθρώπους που δεν μιλούν τη γλώσσα που υποτίθεται ότι κατανοούν και επίσης ορισμένες φορές ε, επιτείνεται η κατάσταση ε, διότι υπάρχουν ετούντε άσυλο που ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα σε κάποιο τμήμα ή σε όλη τη διαδικασία. Ορισμένες φορές λοιπόν οι περισσότεροι είναι απομονεμένοι από τα περισσότερα αν όχι και όλα τα δικαιώματα που έχουν τι επίπεδο πρόσβαση υπάρχει στα κέντρα προσφύγων από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και του δικηγόρου. Μπορεί να γνωρίζει ένα κρατούμενο, να γνωρίζει και να απασχολήσει, να προσλάβει ε, κάποιο νομικό σύμβουλο. Ε, πώς μπορεί ένας αγρόματο κρατούμενος ομαλό ή μια αυγανή γυναίκα ή ανήλικο, ανήλικος να ε, συμπληρώσει τα απαραίτητα έντυπα με τι προθεσμίε που καθορίζονται για να μπορέσουν να γίνουν αποδεκτοί. Υπάρχουν κάποιες ε, αποφάσεις οι οποίες αξιολογούν την ηλικία, κάποιες που καθορίζουν ε, ή αρνούνται το γεγονός ότι ένα άτομο μπορεί να θεωρείται ευάλωτο ε, και αυτές λαμβάνονται από κυβερνητικές και διοικητικές αρχές που δεν είναι βέβαιο ότι γνωρίζουν πολύ καλά τη δουλειά τους ή είναι απόλυτα εξειδικευμένοι γι' αυτό το λόγο. Και επίσης είναι προφανές ότι πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν δικαίωμα για να ζητήσουν έφεση ή προσφυγή για ένα δικαίωμα το οποίο διαθέτουν και δεν το γνωρίζουν. Η τρέχουσα διαδικασία για τις οδηγίες δεν δίνει πολλά στοιχεία υποστήριξης και δίνει μεγάλη διακριτική ευχαίρεια στις κρατικές αρχές, διακριτική ευχαίρεση που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα για την πρόσβαση στην διαδικασία έφεσης και διαπιστώνουμε ότι οι πρωτόδικες αποφάσεις ε, και τα δικαιώματά τους από εκεί και πέρα πρέπει να δίνονται σε μια γλώσσα που να μπορούν να καταλάβουν οι αιτούντες άσελοι. Η πρόσβαση στην τεκμηρίωση και πάλι υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάποιων ε, και αυτό φυσικά μπορεί να έχει και επιπτώσεις στις ε, προθεσμίες προσφυγών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πρόσβαση ε, επί ίσης όρης στην τεκμηρίωση που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών για τη χώρα καταγωγής ε, και ε, στοιχεία από ειδικού όσον αφορά την εγκυρότητα των ταξιδιωτικών τους εγγράφων, παραδείγματα. Ένας κάνει αίτηση ασύλου και από εκεί και πέρα ε, καταθέτει έφεση μετά από την άρνηση της διαδικασίας, ε, θα πρέπει να γνωρίζει όλες τις πληροφορίες. Οποιαδήποτε διατύπωση της διαδικασίας κατάθεσης έφεσης που κατά κάποιο τρόπο αρνείται ε, το δικαίωμα στην προστασία ε, ε ελοχεύει ο κίνδυνος να εκθέσει τον ετούντα άσολα σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως το φοβάται. Υπάρχει και η διάσημη υπόθεση MSS που έριξε κάποιο φως στο γεγονός ότι δεν ήταν αποτελεσματικό το τρέχον σύστημα έφεσης και ε, ο MSS εκτέθηκε σε συμπεριφορά η οποία ήταν αντίθετη στη Σύμβαση ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι προφανές ότι ε, το δικαίωμα της έφεσης βάσει του διπλίνου 2 δεν είναι αυτόματη, αλλά είναι στα χέρια του δικαστηρίου ή της αρμόδιας αρχής που λαμβάνει την έφεση και ορισμένες φορές κατά την άποψή μας θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη μπορεί να μην συμπεριφέρονται στους αιτήτες άσυλο με βάση τα ε, πιο βασικά ε, κριτήρια και τις πιο βασικές αρχές και φυσικά εδώ θα πρέπει να θέσουμε το ίδιο ερώτημα που τέθηκε και νωρίτερα. Πώς μπορεί κάποιος ο οποίος περιμένει επιστροφή βάση του Δουβλίνου να είναι ενήμερος ότι μπορεί να εφεσιβάλει την απόφαση. Είναι δυνατόν ε, να ε, εντοπίσουν κάποιο δικηγόρο, κάποιο νομικό, ο οποίος θα θέλει να τους βοηθήσει και να, τους, ε, και να ξεκινήσει τις προκαταρκτικές διαδικασίες. Μπορεί κάποιοι να κρατούνται σε αεροδρόμια ή σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές όσο εκρεμεί η επιστροφή τους. Πώς μπορούν να λαμβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες. Θα σας ε, παρουσιάσω ένα σύντομο κατάλογο από διάφορες εκδοχές ε, που μπορούμε να έχουμε ε, όταν οι ετούντες ίσολο βρίσκονται αντιμέτωποι με τις διοικητικές διαδικασίες. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίζουμε ότι υπάρχει το δικαίωμα στην αποτελεσματική προσφυγή σε όλες αυτές τις περιπτώσεις και επίσης το, η πρόσβαση σε αποτελεσματική προσφυγή ε, μπορεί να έχει σχέση και με την επανένωση των οικογενειών ή ε, πρόσβαση σε γενικές γραμμές, σε πολιτικά, ε, αστικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα δικαιώματα. Σε ένα λεπτάκι ολοκληρώνω. Το σκεπτικό μου όμω δεν είναι να σα δώσω μόνο ένα κατάλογο, αλλά να δω και τι πιθανέ απαντήσει, απαντήσει από πλευρά ε, των ανθρώπων που δουλεύουν επί τόπου ε, και από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Μα ενδιαφέρουν τα βασικά κριτήρια που αναφέρθηκαν όσον αφορά τον ορισμό μιας αποτελεσματικής προσφυγής, ε, ποια είναι αποτελεσματική, ποια είναι πρακτική και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχουν και κάποια οριζόντια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αναφέρονται. Και εδώ έχω τι τρει τελευταίε μου παρατηρήσει. Με ευφυή χρήση των υφιστάμενων των μηχανισμών χρηματοδότησης και μέσω των εταιρικών σχέσεων με μη κυβερνητικέ οργανώσεις κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία δικαιολογία στο να μην δίνονται πληροφορίες που να είναι σαφείς και στη γλώσσα των ετούντων άσυλων. Ε, οι νομικοί και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει που προσφέρουν συνδρομή στου ετούντε άσυλο θα πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση στου ετούντε άσυλο και σε όλο το υλικό που αφορά τον καθορισμό τη κατάστασή του. Και τέλο, όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι για να λαμβάνουν και να ε, εξετάζουν τις εφέσεις, είτε είναι δικαστικό ή μη δικαστικό, ε, ε, σχεδόν δικαστικό πλαίσιο, θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη τεχνική εμπειρογνωσύνη που είναι απαραίτητη για να διεξάγουν τα καθήκοντά τους. Και φυσικά οι προσπάθειες της ΕΑΣΟ θα πρέπει να είναι πολύ σημαντικές, όπως επίσης και το European Asylum Curriculum. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά το τέλος ε, της ε, συνεδρίασης ενδεχομένως θα έχουμε χρόνο για ανταλλαγή απόψεων, ερωτήσεων κτλ. Χωρίς αργοπορία θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντεν Χέγερ, ο οποίος ε, θα ασχοληθεί με τα ζητήματα στα σύνορα, σύλληψη στα σύνορα κτλ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ ε, για την ε, ε, πρόσκληση. Έχω και μία παρουσίαση PowerPoint. Δεν ξέρω πού ακριβώς προβάλλεται. Ωραία. Θα μιλήσω για ένα λίγο διαφορετικό ζήτημα, το οποίο όμως αφορά στην πρόσβαση προς τη διαδικασία αίτησης ασύλου σε σχέση και με τον έλεγχο των θαλασσίων συνόρων. σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. και κυρίως ε, βεβαίως να δούμε ε, κατά πόσον ο έλεγχος συνόρων και οι αρχές του ασύλου εφαρμόζονται ε, και στους ελέγχους των θαλασσίων συνόρων. Υπήρξαν κάποιες ε, πρόσφατες εξελίξεις. Πέρσι ε, γιναν ε, δεκτές από το Συμβούλιο οι ναυτικές επιχειρήσεις στα πλαίσια της Frontex και επίσης ε, υπάρχει και η συνέχεια της ε, τιμωρίας ε, της απόφασης του δικαστηρίου Τζιράνα, καθώς επίσης και οι τροποποιήσεις του κώδικα Σέγγεν όσον αφορά τα σύνορα. Και επίσης ένα τελευταίο σημείο ε, που θα ήθελα να θίξω είναι ότι δεν είναι τόσο περίπλοκο από άποψη όσο ε, για τον ε, Ευρωπαίο νομοθέτη να αντιμετωπίσει μερικά τουλάχιστον από αυτά τα ζητήματα και εν πάση περιπτώσει εδώ δίδεται μια εξαιρετική ευκαιρία να το πράξει και επομένως να αναλάβει δράση. Γιατί ακριβώς μιλάω και ποια είναι κατά την άποψή μου τα κεντρικά σημεία. Ε, το, προς, το πρώτο θέμα είναι οι διαδικασίες, ποιες είναι οι, ε, ποια είναι τα εχέγγυα τα οποία ε, δίδονται όσον αφορά τον έλεγχο στα σύνορα, διαφάνεια κτλ. Έχουμε την ε, περίπτωση ε, των ε, επικριτικών εκθέσεων CPT όσον αφορά το θέμα της Ιταλίας και της βίαιης απόθεσης προσφύγων από την χώρα αυτή. Για την υπόθεση αυτή αναμένουμε και την απόφαση του δικαστηρίου. Το 2008 ε, και το 2009 υπήρξαν ε, επαναπροωθήσεις από την Ιταλία προς την Τινησία και την Λιβύη που σταμάτησαν βεβαίως λόγω των γεγονότων της προηγούμενης ε, άνοιξης. Πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι συμφωνίες με τις αφρικανικές χώρες οι οποίες είναι μυστικές εκτός από μια συμφωνία ανάμεσα στην Ισπανία και το πράσινο ακροτήρι. Ε, θα πρέπει από τη στιγμή που ο έλεγχος των ε, συνόρων αποτελεί ε, στοιχείο της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι δυνατόν οι συμφωνίες με τρίτες χώρες να παραμένουν μυστικές. Θα ήθελα πρώτα να αναφερθώ στις ε, διαδικασίες και πώς ε, το Συμβούλιο αποφάσισε να λύσει ε, το ζήτημα της ετύχης που θα πρέπει να έχουν τα πλοιάρια τα οποία σταματώνται στη θάλασσα. Ε, το θέμα αυτό βρίσκεται εγκρεμή ενώπιον του δικαστηρίου και θα υπάρξει απόφαση ε, μέσα στον επόμενο χρόνο. Ε, το σημαντικό είναι να γίνει σεβαστή η αρχή της μη επανεκτόπισης των non-refoulement. Ε, και βεβαίως ε, σύμφωνα και με τα όσα γράφω και στο γράφημά μου εδώ ε, μπορούν να υπάρξουν ανακρίσεις, να γίνουν ανακρίσεις ε, τόπου και στους επιβαίνοντες στα πλοία και επομένως ενδεχομένως να ληφθεί η απόφαση να να επαναπροωθηθούν στη χώρα από την οποία να προέρχονται. Η απόφαση ε, του ε, Συμβουλίου που εφαρμόζει και τον ε, κώδικα Σέγγεν οπωσδήποτε διασφαλίζει κάποια εχέγγυα όσον αφορά τη διαδικασία αλλά επιτρέπει την απαγόρευση εισόδου. Και πρέπει να πω ότι έτσι όπως διατυπώνονται τα πράγματα, ε, στην ουσία πρόκειται για μια δημιουργική αντιμετώπιση του νόμου κατά την ε, άποψή μου. Ε, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει το δικαστήριο όταν θα βγάλει την απόφασή του, αλλά όταν ε, στέλνεις ανθρώπους ε, πίσω στη χώρα από την οποία ε, προελθούν στην ουσία είναι ε, απαγόρευση εισόδου και επομένως οι ανακρίσεις δεν γίνονται με διαφανή τρόπο αλλά γίνονται με συγκεκριμένο σκοπό που είναι ακριβώς είτε η σύλληψη, είναι η σύλληψη των ανθρώπων και επομένως να, τους, να επιστρέψουν τους ανθρώπους αυτούς στις χώρες από τις οποίες προήλθαν λαμβάνοντας υπόψη και εφαρμόζοντας πλήρως τον κώδικα εξωτερικών συνόρων το Σέγγεν. Οδηγούμε στην πρώτη μου σύσταση λοιπόν ή μάλλον ερώτηση θα μπορούσα να πω. Ε, ερώτηση λοιπόν, οι <coughs> επιχειρήσεις ε, ε, του ελέγχου των θαλασσίων ε, συνόρων μπορούν να θεωρηθούν υπό τον, Ευρωπαϊ... Ενωσιακό Νόμο ως επιτήρηση των συνόρων και επομένως να διέπονται από όλες τις εγγυημένες διαδικασίες. αυτά που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή άρνηση εισόδου, ανακρίσεις επιτόπου κτλ. Δεύτερη σύσταση σχετίζεται με την μυστικότητα των συμφωνιών ε, η Ισπανία έχει κάνει 6-7 συμφωνίες με αφρικανικές χώρες, η Ιταλία έχει κάνει ε, διάφορα πρωτόκολλα συμφωνίας ε, με την Λιβύη. Και επίσης πρέπει να πω ότι σχετικά με την Ιταλία και μετά τα γνωστά ατυχήματα και τις ατυχείς καταστάσεις που διαμορφώθηκαν με τους τιμήσιους μετανάστες στην Ιταλία υπήρξε μια αναθεώρηση της συμφωνίας την 5η Απριλίου του 2011. Παρ' όλα αυτά ε, υποχρεούται η Τινησία να... Ε, ε, οι Ιταλοί επαναπροωθούν τους Τινησίους στη χώρα τους και η Τινησία πρέπει να τους υποδεχτεί. Και αυτό εάν ξεπεραστεί ο αριθμ, ένας αριθμός και ένα συγκεκριμένο ποσοστό ατόμων ή σκαφών υπάρχουν και οι συμφωνίες ανάμεσα στην Ισπανία και τις αφρικανικές χώρες που ανέφερα προηγουμένως και ε, υπάρχει όσον αφορά την περίπτωση της Ισπανίας κάποιος έλεγχος Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπάρχει βέβαια και μια νέα ρήτρα η οποία λέει ότι θα πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες, όλα τα ε, ε, σημεία διάβασης ε, κοινών συνόρων και όλες οι συμφωνίες οι οποίες διέπουν το, τα, σημεία περάσματα κοινών συνόρων. Όλες λοιπόν οι αποφάσεις οι οποίες σχετίζονται και οι συμφωνίες που σχετίζονται με αυτό θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Κομισιόν έστω και αν εμπίπτουν σε διμερή διμερείς ε, συμφωνίες ε, των χωρών. Οτιδήποτε λοιπόν αφορά την ε, επίβλεψη των συνόρων, οτιδήποτε αφορά τον έλεγχο των συνόρων και οποιασδήποτε συμφωνίες γίνονται από αυτού του θέματος θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και με τον τρόπο αυτό ενδεχομένως θα δοθεί περισσότερη δυνατότητα ελέγχου καθώς επίσης και διαφάνεια στην όλη διαδικασία. Ε, σας έχουμε, έρωσουμε, δεν είχαμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, σας έχουμε ε, όλα τα στοιχεία τα οποία θα σας οδηγήσουν στην ιστοσελίδα μας ε, έτσι ώστε να κατανοήσετε πληρέστερα τη δουλειά μας και να δείτε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Πράγματι, σας ευχαριστώ και για τις συστάσεις, τις προτάσεις που έχετε κάνει σε εμά ως νομοθέτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει κάποιος έλεγχος των διμερών αυτών συμφωνιών κάτω μέρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες και επίσης αναφερόμενοι στην ε, παρουσίαση του κυρίου Φάζων είναι πολύ σημαντικό όταν συντάσσουμε νομοθεσία να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα, πώς οι λέξεις, οι φράσεις της νομοθεσίας θα εφαρμοστούν στην πράξη, εάν εφαρμοστούν. <clears throat> Αυτό θα ήθελα να πω και έχετε πέντε λεφτά για να θέσετε ερωτήματα αν θέλετε. Κύριος Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους τέσσερις ομιλητές για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Χέιρ. Βασίζεται το επιχείρημά σας στο ότι κατά τη διάρκεια κάποιας ναυτικής επιχείρησης. Θα πρέπει πάντα και εκεί να υπάρξει εγγύηση της αρχής της μη επαναπρόθεσης. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ότι στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιώματα που έχουν τα άτομα αυτά για παροχή ασύλου θα πρέπει να τύχουν προστασίες. Αυτό το οποίο παραγνωρίζεται είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ακολουθούν παράνομες οδούς εμπλέκεται το θέμα της λαθρεμπορίας ανθρώπων, της εγκληματικότητος. Όταν εσείς σταματήσετε, να αναχαιτήσετε ένα πλοίο, ώστε να δώσετε το δικαίωμα ασύλου σε αυτούς τους ανθρώπους, αν τους φέρετε στην Ευρώπη, εσείς βοηθάτε και υποστηρίζετε ένα κύκλωμα λαθρεμπορίου ανθρώπων. Το ερώτημά μου είναι το εξή Ενώ εγώ κατανοώ και συμφωνώ ότι πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα ασύλου σε οποιοδήποτε το χρειάζεται αυτό. Σίγουρα δεν θα πρέπει να το πράξουμε αυτό με ένα τέτοιο τρόπο που μας καθιστά συνενόχους σε αυτό το οποίο είναι ουσιαστικά μια εγκληματική δραστηριότητα. Είναι κάτι διαφορετικό να έρθει κάποιος στη χώρα μας, στα σύνορα, στο αεροδρόμιο και να ζητήσει άσυλο. Είναι τελείως διαφορετικό το να σταματήσουμε μια δραστηριότητα η οποία είναι μια παράνομη δραστηριότητα, να συλλάβουμε ένα πλοίο και να γίνουμε μετά συνένοχοι σε αυτή τη δραστηριότητα στο όνομα της παροχής ασύλου. Αυτό είναι λοιπόν ένα πολύ λεπτό και δύσκολο θέμα. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μου δώσετε μια απάντηση γι' αυτό. Συμφωνώ με αυτό που λέτε, κύριε Βουλευτά, ότι αυτό είναι ένα τεράστιο δίλημα. Και μιλώ ως, ε, νο, νομικός και όχι σας, ως πολιτικός. Ως νομικός όμως θα σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι είναι θεμητό να κάνετε πράγματα στη θάλασσα, στα θαλάσσια σύνορα, που δεν θα κάνετε σε χερσαία ή σε άλλα σύνορα. Δηλαδή να σταματήσετε κάποιον, να τον ξαναδιώξετε χωρίς να του δώσετε καμία διαδικαστική ε, εγγύηση. Μήπως αυτός είναι ένας τρόπος να παρακάμψετε όλους τους κανόνες που ισχύουν στον κώδικα του Σέγκεν. Μπορεί να σας φανεί τυπική αυτή η απάντηση, αλλά νομίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα ατενίσει έτσι τον κώδικα σύνορων του, της ζώνης του Σέγγεν. Αν πρέπει να έχετε κάποιους κανόνες στα σύνορα και αν αποφασίσετε από μόνο σας να σπρώξετε το σύνορο στη θάλασσα για να μην χρειάζεται να εφαρμόσετε αυτούς τους κανόνες, εγώ ως ε, δικηγόρος, ως νομικός βλέπω να υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Φυσικά υπάρχει το δίλημα αυτό που λέτε αν τα άτομα αυτά θα πρέπει να τα στείλουμε από εκεί που ήρθαν ή αν θα πρέπει να τα φέρουμε σε έδαφο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να, δι, για να υποβληθούν στι προβλέψεις διαδικασίε. Ούτε και εγώ έχω λύση για το δίλημά σα, λοιπόν. Το βλέπω αυτό το θέμα από την πλευρά του ευρωπαϊκού δικαίου και του δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρώ ότι πρέπει τα άτομα αυτά να τύχουν επεξεργασία σε σχέση με την αίτηση ασύλου. Επίση, θα πρέπει να αναφέρουμε, λέει ο κ. Φάλσον, ότι αυτοί οι οποίοι ζητούν άσυλο ακολουθούν πολλές φορές μη κανονικούς δρόμους για να μπουν στα σύνορα μιας ευρωπαϊκής χώρας, όχι μόνο από τη θάλασσα, αλλά και από αεροδρόμια και άλλους τρόπους. Πολλοί λοιπόν έρχονται με αντικανονικό τρόπο και ζητούν άσυλο. Εμείς δεν θέτουμε θέμα του αν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο αυτοί, παρά μόνο σε αυτούς που έρχονται δια της θαλασσίας οδού το ότι οι αιτούντες άσυλο έρχονται με παράνομα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό οφείλεται γιατί υπάρχουν μέτρα τέτοια τα οποία κάνουν σχεδόν αδύνατο να μπορέσει κάποιο να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά από τη Σομαλία. Κάποιο από το Ιράν, από το Αφγανιστάν, από το Ιράκ δεν μπορεί <clears throat> να έρθει νομίμω στο έδαφο τη Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το γεγονό ότι εμεί δεχόμαστε ότι από τη στιγμή που έρχονται και ζητούν άσυλο θα πρέπει να τύχουν νομικής προστασία. Λοιπόν, το να σταματάμε κάποιον στη θάλασσα δεν είναι μια λύση, γιατί ουσιαστικά στέλνετε πίσω κάποιον σε μια χώρα όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα του κινδυνεύουν να τύχουν παραβίασης. Άλλα ερωτήματα, λέει η πρόεδρος. Θέλετε να πείτε κάτι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Αμέσως αρχίζει το επόμενο πάνελ για την επιβολή κυρώσεων. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές και ευχαριστώ όλους αυτούς οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τη συζήτηση. Για να συνεχίσουμε λοιπόν. Στη συνέχεια ε, της συνεδρίασης αυτής που είναι πάρα πολύ σημαντική ε, όπως ήταν και η σημερινή ε, πρωινή συνεδρίαση για να δούμε τα θέματα τα οποία θα οδηγήσουν στο Κοινοβούλιο στις σχέσεις μεταξύ του Συμβουλίου που αυτή τη στιγμή εκπροσωπείται από την Πολωνία και από και ημών των Ευρωβουλευτών ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε γρήγορες λύσεις ε, για τα θέματα του ασύλου. Θα ήθελα να δώσω το λόγο λοιπόν στην κυρία Τίνα Άκετοφ, μου είναι αδύνατο να προφέρω σωστά το όνομά σα, ζητώ συγγνώμη, μέλο τη Επιτροπή Μετανάστευση Προσφύγων και Πληθυσμού τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Παρακαλώ. Grazie. Thank you. Uh, Ευχαριστώ. Άκετοφτ λέγομαι. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο ακόμα και στα σουηδικά να προφέρει κάποιο το όνομά μου. Σας ευγνωμονώ διότι δώσετε τη δυνατότητα στο Συμβούλιο της Ευρώπης ε, να μιλήσει και να συζητήσει για αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα το οποίο μας αφορά όλους. Ε, είτε είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε δεν είμαστε. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί είμαι μέλος ε, μιας ad hoc υποεπιτροπής ε, του Συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης που ασχολείται με τα θέματα άφηξης ε, κράτησης και των συνθήκων κράτησης. Θα επισκεφτούμε τη Λαμπεντούσα και την ε, Τουρκία, έχουμε πάει και στη Μάλτα και στην Ελλάδα, όπως φαντάζομαι ότι θα έχετε κάνει και εσείς. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η αντιμετώπιση του θέματος της κράτησης ε, των ετούντων άσυλη αποτελούσε προτεραιότητα για την Κοινοβουλευτική Συνέλευση εδώ και αρκετά χρόνια και είναι ένα από τα βασικά μας ζητήματα. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπάρχει και σημαντικό ε, αριθμός κανόνων και προτύπων που αφορούν και τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, φυσικά και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει και ένα σύστημα για να εντοπίζονται ελλείψεις, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Επιτροπή Κατά των Βασανισμών, την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ούτω καθεξής η κράτηση παράνομων μεταναστών και τούτον άσυλο έχει αυξηθεί ε, τα τελευταία χρόνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεκαπλασιάστηκαν ε, τα ποσοστά σε σχέση με τη δεκαετία του 90. Στη Γαλλία από 759 άτομα το 2003 έχουμε φτάσει στα 1724 άτομα το 2007 η αύξηση της κράτησης ε, δεν γίνεται μόνο λόγω της αυξημένης ροής μεταναστών και παράνομων μεταναστών και του τον άσυλο, αλλά έχει αυξηθεί και ο αριθμός ε, των αιτίων για τους λόγους αποφασίζεται η κράτηση και είναι και μεγαλύτερος ο χρόνος κράτησης. Και η οδηγία έχει διευκολύνει την κατάσταση με το όριο 6 μηνών, το οποίο παρατείνεται στους 18 μήνες σε κάποιες περιπτώσεις και δυστυχώς αυτό έχει αποστείλει το μήνυμα στα κράτη-μέλη ότι η μακροχρόνια παρόμοιες κρατήσεις είναι αποδεκτές. Κάποιες φορές ε, ως πολιτικοί έχουμε την τάση να περιπλάκουμε κάποια θέματα. Ε, όταν ε, στην πραγματικότητα το μόνο το οποίο πρέπει να αναρωτηθούμε είναι κατά πόσον είναι απαραίτητο να κρατούνται τόσοι πολλοί άνθρωποι και αν όντω πρέπει να κρατούνται, αν πρέπει να κρατούνται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Η απάντηση θα πρέπει να είναι απλή. Αλλά ακόμα και το σημείο κίνησης στο διεθνέ δίκαιο είναι σαφέ. Η κράτηση θα πρέπει να είναι η τελευταία λύση. Όχι η πρώτη, ούτε καν η δεύτερη, αλλά η έσχατη. Και όσον αφορά την ε, σύμβαση των προσφύγων, η κράτηση των ετούντων άσφυλων δεν θα γίνεται μόνο και μόνο επειδή καταθέτουν μια αίτηση ή γιατί έχουν εισέλθει παρανόμω σε μια χώρα. Και δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι οι κρατούμενοι μετανάστες δεν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα. Ε, πολλές φορές κρατούνται σε συνθήκες οι οποίες είναι απάνθρωπες και είναι και χειρότερες από αυτές που επιφυλάσσουμε στις εγκληματίες. Μετά από αυτή την εισαγωγή λοιπόν κυρίες και κύριοι θα ήθελα να σας δώσω τρεις αρχές κράτησης ε, που προκύπτουν από τα ψηφίσματα της κοινοβουλευτική Συνέλευσης για την κράτηση των παρανόμων μεταναστών και των ετούντων άσυλο στην Ευρώπη και ελπίζουμε να βοηθήσουν στη συζήτηση για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη συζήτηση του ζητήματος. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η κράτηση θα πρέπει να είναι η έσχατη λύση. Θα πρέπει να αναζητήσουμε άλλες λύσεις πριν αποφασίσουμε ότι η πλέον κατάλληλη λύση είναι η κράτηση. Δεύτερον, εάν αποφασιστεί το θέμα της κράτησης, θα πρέπει να συνάδει με το διεθνές δίκαιο, που περιορίζει τους ε, τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιείται ε, η κράτηση. Χρειάζεται φυσικά μεγαλύτερη σαφήνεια για το θέμα αυτό, το γνωρίζω, αλλά όταν διατάσσεται η κράτηση θα πρέπει να γίνεται κράτηση σε κατάλληλες συνθήκες, με κατάλληλες δραστηριότητες και υποστήριξη. Ελπίζω οι υπόλοιποι ομιλητέ να εμβαθύνουν στο θέμα των εναλλακτικών λύσεων τη κράτηση, ακόμα και αν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διευκρινίσουμε και να εξετάσουμε περαιτέρω. Θα ήθελα όμω να πω κάποια από τα προφανή αίτια για τα οποία χρειαζόμαστε εναλλακτικέ λύσει. Καταρχά υπάρχει ε, το χρηματοοικονομικό κομμάτι. Είναι φτηνότερες οι εναλλακτικέ λύσεις. Στον Καναδά ένα πρόγραμμα κράτησης στοιχίζει 12 με 15 καναδικά δολάρια την ημέρα, ενώ μια αντίστοιχη εναλλακτική λύση είναι πολύ φθηνότερη, είναι στα 5 δολάρια την ημέρα, αλλά είναι το ανθρώπινο κόστος το πιο σημαντικό από το οικονομικό. Υπάρχουν σημαντικές ε, ψυχολογικές συνέπειες που ορισμένες φορές είναι δυσβάσταχτες. Ο Σουηδί θα πρέπει να επισημάνω ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης αναφέρεται κυρίως στο γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις ε, στην κράτηση, αλλά αυτές είναι εναλλακτικέ ε, λύσεις στη φυλάκιση και δεν έχουν σχέση με τους ετούντες άσυλο και τους παράνομους μετανάστες. Και συγγνώμη που επαναλαμβάνω συνέχεια το ίδιο πράγμα, αλλά φαίνεται ότι ευνοούμε λιγότερο ανθρώπους που δεν έχουν διαγράψει κανένα δίκημα, αλλά προς προσπαθούν να έρθουν σε μια άλλη χώρα για να κερδίσουν τα προστοζήν. Εάν όμως εξετάζουμε το θέμα της κράταση, θα πρέπει να γίνεται βάση διεθνού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα ε, Δικαιώματα ε, βοηθά μεν, αλλά δεν αποτελεί πανάκια και χρειάζεται φυσικά καλύτερη ο συντονισμό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η κράτηση λοιπόν μόνο για την ε, παράνομη κρά, είσοδο και ε, απέλασης. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε είναι ότι ένα από τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Χάρτα είναι ότι για να είναι νόμιμη η κράτηση θα πρέπει να είναι απαραίτητη. Παραδείγματο χάρη, κάποιο ο οποίο δεν αποτελεί καμία απειλή για κάποιον. Έχει στέγαση, έχει χρηματοδότηση και όλε τι απαραίτητε διασφαλίσει. Μπορεί επί τη αρχή να τελή υποκράτηση αν τηρούνται άλλε προποθέσει τη συνθήκη. Παραδείγματο χάρη ε, κράτηση εν ώψη απέλαση. Και θα πρέπει να πω ότι δυστυχώ ακόμα και η ίδια μου η χώρα το χρησιμοποιεί αυτό ω αιτιολογία. Για να κατανοήσουμε πλήρως ε, τους περιορισμούς ε, της κατάστασης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των διεθνών νομικών μέσων. Το 2004 και το 2005 είχαμε το περιθώριο να μιλάμε για ε, μη αναμενόμενες αφέξεις παράνομων μετανοστών και του Ντονάσολο σήμερα γνωρίζουμε ότι αναμένουμε την άφηξη αυτών των ανθρώπων. Ήταν αλήθεια ότι δεν περιμέναμε την Αραβική Άνοιξη και τις αφήξεις από την ε, Βόρεια Αφρική, αλλά ε, οι αριθμοί των ανθρώπων που καταφτάνουν δεν είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους μετανάστες που υποδεχόμασταν προηγουμένως. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες υποδοχής ε, και αν υπάρχουν ε, κέντρα κράτησης θα πρέπει να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και την κατάλληλη υποδομή. Η οδηγία για τις επιστροφές έχει προϋποθέσεις ε, για τα θέματα κράτησης και το ίδιο έχουμε και στις κατευθυντήρες γραμμές για τις ε, καταναγκαστικές επιστροφές. Αλλά θα πρέπει ε, ε, να γνωρίζουμε και τι ακριβώς ε, γίνεται στις συνθήκες κράτησης. Γι' αυτό και εμείς ε, στη συνέλευση έχουμε τα 15 ελάχιστα πρότυπα για τις συνθήκες κράτησης των παράνομων μεταναστών και των ετούντων άσυλων και ζητήσαμε να ετοιμαστούν και ευρωπαϊκοί κανόνες για την κράτηση των ανθρώπων αυτών. Αυτό θα συμπληρώσει και τους ε, παρόντες ευρωπαϊκούς κανόνες που είναι και μία από τις μεγαλύτερες συνεισφορές που έχει κάνει το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τομέα αυτό μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, ε, καταπολέμηση των βασανισμών. Να συνοψίσω ως πολιτικός της χώρας μου στην Ευρώπη και ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης ζητώ την κατανόησή σας αν επαναλαμβάνω συνεχώς τα ίδια πράγματα κράτηση θα πρέπει να έχουμε μόνον όταν είναι απαραίτητη. Θα πρέπει να υπάρχει αλληλοκατανόηση ως πρωτο, στο τι ακριβώς εννοούμε απαραίτητο. Η κράτηση θα πρέπει να είναι ανάλογη με το στόχο που προσπαθούμε να επιτύχουμε και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ιδέουσα ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος της ελευθερίας του ατόμου και του ε, συμφέροντος του κράτους. Και ε, βάσει αυτών των δύο στόχων, χωρίς να λέω ότι η αυτόματη υποχρεωτική κράτηση παραβιάζει και τις δύο αυτές αρχές. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να βρούμε ποιες είναι οι εναλλακτικέ λύσεις για την κράτηση. Αλλά εάν κρατούμε ανθρώπους ε, για λόγους μετανάστευσης, θα πρέπει να ζουν υπό ανθρώπινες συνθήκες και δεν κρατούνται άνθρωποι που θα έπρεπε να είναι ελεύθεροι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Μας χαροποιεί πάρα πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακούμε αυτά τα οποία ακούσαμε από εσά, γιατί είναι προφανές, είναι απόλυτα κατάδειλο ότι δεν μπορούμε να συλλαμβάνουμε και να κρατούμε κάποιον ο οποίος αγωνίζεται για την ελευθερία και έρχεται στην Ευρώπη και το πρώτο πράγμα που γίνεται του βάζουν χειροπέδες και τον βάζουν σε ένα κελί. Αυτό δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τις ευρωπαϊκές αρχές και χαίρομαι που κι εσείς στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχετε αυτή την άποψη και μπορείτε να το επαναλάβετε σήμερα. Είναι επίσης πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπατε, η ανάγκη να αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις. Πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις έναντι της κράτησης και μπορεί να είναι πιο φτηνές. Και εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούμε να πείσουμε τις ε, ε, εθνικές κυβερνήσεις να αφήσουμε τους ανθρώπους ελεύθερους και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να είναι στην αγορά εργασία. Ότι αυτό είναι πολύ πιο απλό και φθηνό από το να του έχουμε στη φυλακή. Χαίρομαι λοιπόν που το αναφέρατε το θέμα αυτό. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Χιλ Μπάθο Μαρία Τερέσα, η οποία είναι διευθύντρια του, των μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο, νομικών μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Νιουκάσλ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα κυρίε και κύριοι. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που μπορώ και πάλι να λάβω το λόγο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με διαφορετική ιδιότητα και σε μια στιγμή που το Κοινοβούλιο έχει ήδη ενσωματώσει την εφαρμογή της Συνθήκης Λισαβόνας και έχει τις νομοθετικές εξουσίες που θεωρούμε όλοι ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να χρησιμοποιήσουμε ένα πιο προορατικό τρόπο από ό,τι έχει πράξει στο παρελθόν με τις δυνατότητες που είχε στο παρελθόν πριν από την θέση εφαρμογή της Λισαβόνας. Στην παρουσίασή μου θα αντιμετωπίσω μία σειρά συγκεκριμένων θεμάτων. Δεν θα πω τώρα στις λεπτομέρειες της πρότασης αναδιατύπωσης των ρητρών και διατάξεων που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολλά έγγραφα τα οποία έχουν υποβλεθεί και από την Amnesty International και από την ύπατη αρμοστία για του πρόσφυγε και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για του Προσφύγε που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αυτά λεπτομεριακά. Εγώ θα εστιάσω σε μία σειρά από συγκεκριμένα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να αναφερθώ στις γενικές αρχές οι οποίες έχουν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως τι αυτές θα πρέπει να διέπουν πάντα την νομοθετική ατζέντα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια θα εστιάσω σε ορισμένε από αυτέ τι αρχέ, όπω έχουν καταγραφεί στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εστιάσω ιδιαίτερα λοιπόν στο δικαίωμα ασύλου. και θα αναπτύξω κάποια επιχειρήματα σε σχέση με την ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που δεν έχει ίσως τύχει επαρκούς προσοχής. Θα σταθώ λιγάκι επίσης και στο παράγωγο δίκαιο και τα διδάγματα τα οποία έχουμε, ε, μπορούμε να αντλήσουμε και τα οποία μπορούν να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τα εκκρεμή θέματα ενώπιών μας. Πρέπει να ξεκινήσω τονίζοντας κάτι το οποίο έχει ήδη λεχθεί σε διάφορες παρεμβάσεις. Συζητούμε θέματα διοικητικής κράτησης κράτησης ατόμων τα οποία καταρχήν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν το άσυλο και ατόμων οι οποίοι μπορεί να είναι πρόσφυγες ακόμα και αν δεν έχουν τύχη αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε στις αρχές και τις υποχρεώσεις του διεθνούς που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να δράσουν με έναν τρόπο. Δεν μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν διαπράξει αδικήματα ή τα οποία περιμένουν την δίωξή του, την ε, δίκη του και τη δίωξή του βάσει του ποινικού δικαίου. Οι δύο βασικέ αρχέ οι οποίε διέπουν τα θέματα αυτά είναι το άρθρο 6 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όπου αναφέρεται το δικαίωμα όλων στην ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια και επίσης το άρθρο αυτό δεν έχει ακόμα αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητες του και περιμένουμε να ακούσουμε και την απόψη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε σχέση με το περιεχόμενό του. Αυτό είναι το άρθρο 18 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ασύλου. Λέει ότι το δικαίωμα στο άσυλο θα πρέπει να τύχει εγγύησεως στο φως της Σύμβασης της Γενέβης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων και των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μας λέει λοιπόν αυτή η χάρτα. Λέει ότι βάσει του άρθρου, η σύμβαση της Γενέβης, ότι βάσει του άρθρου 31 σύμβαση της Γενέβης δεν πρέπει να εφαρμόζονται κυρώσει τους πρόσφυγες λόγω της παράνομης εισόδου ή παρουσίας τους στο έδαφος ενός κράτους ή αυτών που είναι παρόντες χωρίς άδεια στο έδαφος και την επικράτεια μιας χώρας. Μας λέει επίσης ότι δεν μπορούν να επιβληθούν περιορισμοί στην κίνηση αυτών των ατόμων πέραν αυτών που είναι απαραίτητες και μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητες μέχρι ότου το καθεστώς τους στη χώρα αυτή ή η είσοδός τους σε μια άλλη χώρα έχει συμπληρωθεί. Επομένως αυτά βρίσκονται μέσα στη σύμβαση της Γενέβης η οποία διέπει το περιεχόμενο του άρθρου 18. Το άνθρωπο αυτό για το άσυλο αναφέρεται στο δικαίωμα να ζητήσει κανεί άσυλο, αλλά προχωρά και πολύ περισσότερα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει κληθεί να δώσει μία απάντηση στα θέματα αυτά και περιμένουμε ακόμα μία γνωμοδότηση για τα θέματα αυτά. Δυστυχώς η πρόταση του Γενικού Εισαγγελία δεν αναφέρεται στο περιεχόμενο του άρθρου 18 και δεν απαντά το ερώτημα που έθεσε ένα ακυρωτικό δικαστήριο σε σχέση με την εμβέλεια του άρθρου 18 και μέχρι ποιου βαθμού μπορούν να εκταθούν οι εγγυήσει που βασίζονται στο άρθρο αυτό στην Χάρτα Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά σε σχέση με το περιεχόμενό του, οποιαδήποτε εξαίρεση από το άρθρο 18 βάσει τη νομοθεσία Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνάδουν με τι βασικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ αναφέρεται η αρχή τη αναλογικότητα, η αρχή τη αναγκαιότητα, το δικαίωμα σε χρηστή διοίκηση και ασφάλεια δικαίου που πολλές φορές οδηγούν σε πιο εκτενείς εγγυήσεις, το δικαίωμα αποτελεσματικής θεραπείας και η αρχή της αποκατάσταση. Δηλαδή η υποχρέωση στις αρχές να αποκαταστήσουν τις ζημίες οι οποίες προέρχονται από μία, παραδείγματος χάρη, μη ε, νόμιμη κράτηση. Έχουμε επίσης την παράγωγη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναφέρεται στη νομική βάση κράτησης και τις συνθήκες που πρέπει να πληρεί η κράτηση για να είναι νόμιμη. Σε σχέση με την νομική βάση, η ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται στη στιγμή που γίνεται η προσπάθεια, μπαίνει κάποιος να, στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν κρατείται πριν καταθέσει την αίτηση ασύλου και στην στιγμή που αφορά υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει αποφασιστεί να απελαθεί. Τα άτομα τα οποία θα απελαθούν δεν έχουν δικαίωμα να μείνουν σε μια χώρα και επομένως δεν μπορούν να απολαμβάνουν προστασίας βάση του διεθνούς δικαίου. Αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα στην πράξη. Άτομα τα οποία αναμένουν να απελαθούν μπορεί να περιμένουν να απελαθούν ή να μεταφερθούν σε άλλη χώρα βάσει τον κανονισμό του Δουβλίνου, επομένω η περίπτωσή του δεν έχει εξεταστεί, δεν έχει εκδικαστεί πλέον. Μπορούν να μεταφερθούν κάπου αλλού με βάση τη αρχή τη ασφαλέστερη χώρα ή βάσει διεθνού νομοθεσία η οποία επιβάλλει ένα δικαίωμα ένσταση, προσφυγή καλύτερα, από το εξωτερικό μια χώρα. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα αυτά που βρίσκονται σε αυτές τις καταστάσεις μπορεί πράγματι να είναι πρόσφυγες των οποίων η υπόθεση δεν έχει ακόμα εκδικαστεί και επομένως το καθεστώς τους ως προσφύγων δεν έχει τύχει αναγνώρισης. Στην περίπτωση αυτή η οδηγία 2004 αναφέρει μία σειρά από ελάχιστα πρότυπα. Το Κοινοβούλιο στην περίπτωση αυτή έχει δυνατότητα να αντλήσει κάποια συμπεράσματα από αυτή την οδηγία σε σχέση με την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην περίπτωση ΚΑΤΣΟΕΦ έχει ήδη αντιμετωπίσει το θέμα της νομιμότητας της κράτησης. Και, αυτή η κράτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια λογική πιθανότητα ε, μεταγωγής, μετακίνησης του κρατουμένου. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η προοπτική ε, ότι θα μεταφερθεί ο κρατούμενος, πρέπει να απελευθερωθεί αμέσως. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν μπορεί να αντλήσει από, αυτή την υπόθεση διδάγματα ώστε να προχωρήσει σε περισσότερες διασφαλίσεις και να έχει περισσότερες λεπτομέρειες στην οδηγία περί υποδοχής. Ένα τελευταίο στοιχείο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ότι το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγγνώμη, έχει αναπτύξει μια νομολογία όπου όλο και περισσότερο επιμένει στις υποχρεώσεις των κρατών μελών και ιδίως στις θετικές <clears throat> υποχρεώσεις και όχι μονάχα τις αρνητικές υποχρεώσεις, δηλαδή να μην πάρει μέτρα σε βάρος των κρατουμένων. Οι θετικές υποχρεώσεις μπορεί να σημαίνουν την ανάγκη να τροποποιηθεί η εθνική ε, νομοθεσία όπως έγινε στην, ε, σε μια περίπτωση που ενέπλεκε την Βουλγαρία και ΑΟΑΤ εναντίον Βουλγαρίας και επίσης είναι σαφές το, σαφής η υποχρέωση τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε κράτηση να μην εμποδίζονται να ασκήσουν αποτελεσματικές διαδικασίες για να καθοριστεί το καθεστώς τους. Και επίσης κάτι το οποίο συζητήθηκε στην προηγούμενη, στο προηγούμενο πάνελ είναι το θέμα του πώς τα κράτη-μέλη αρνούνται την εφαρμογή της γενικής αρχής του κοινοτικού δικαίου σε ενέργειες αναχέτησης πλοίων στην ανοιχτή θάλασσα, στα πλαίσια συνεργασία με τρίτες χώρες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χιλμπάθο. Συγγνώμη, αλλά εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάμε για 2, 3, 4 λεπτά το πολύ. Και έχουμε το πρόβλημα της διερμηνίας, έχουμε το πρόβλημα των ανθρώπων, του αθμού, των αυτών οι οποίοι παρεμβαίνουν. Ενώ σε ένα δικαστήριο ή σε ένα πανεπιστήμιο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γι' αυτό λειτουργούμε έτσι, δύσκολο να το αλλάξουμε σήμερα αφού δεν μπορούμε να αλλάξουμε όλο το δίκαιο του ασύλου, ίσως μπορούμε να αλλάξουμε κάτι σε αυτά τα πράγματα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Φιλίπ Αμαράλ, τον οποίο γνωρίζουμε. Είναι γνωστός για την προσήλωσή του στον αγώνα υπέρ των προσφύγων και του δίνω το λόγο αμέσως. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την πρόσκληση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών που με κάλεσε για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, τελευταίες μελέτες που κάναμε όσον αφορά ε, τους ε, τρόπους κράτησης και τις απόψεις που έχουμε όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής. Ε, και αν έχω χρόνο θα μιλήσω, θα αναφερθώ και σε κάποιες εναλλακτικέ προτάσεις. Είναι ενδιαφέρουσε οι εναλλακτικέ προτάσεις, λέει ο Πρόεδρο, να το κάνετε. Η αποστολή το, υπηρεσία της υπηρεσίας ε, προσφύγων των Ιουσιτών ε, είναι να συνοδεύει, να υπηρετεί και να δίνει νομικής, νομικές συμβουλές ε, σε ε, πρόσφυγες, ε, καθώς επίσης και άτομα που υποχρεούνται να μεταναστεύσουν. Επί σειρά ετών έχουν γίνει επισκέψεις σε κέντρα κράτησης, έτσι ώστε να δούμε αν υπήρχε, υπήρχε, τρόπος να δούμε ποια είναι τα άτομα που είναι πιο ευάλωτα και πιο, ε, ε, πιο αυτά που χρειάζονται με περισσότερη ανάγκη και που είναι πιο ευάλωτα. Ε, επομένως εμείς ήρθαμε σε επαφή και υποβάλαμε συνεντεύξεις σε 685 κρατούμενους που ζητούν άσυλο, καθώς επίσης και μετανάστες χωρί ταξιδιωτικά έγγραφα από 21 χώρε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 10 έως 64 ετών. Εμεί βασιστήκαμε σε μια σειρά σταθερών ε, παραγόντων αλλά και μεταβλητών που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις και συγκεκριμένα άτομα. Ε, όμως ε, βλέπουμε ότι ε, το κατά πόσο είναι ευάλωτο ένα άτομο ε, εξαρτάται και από τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο πρόσφυγας βλέπει τον εαυτό του και από τι προσπαθεί να κρυφτεί. Είδαμε ε, λοιπόν ότι υπάρχουν τα άτομα τα οποία είναι σαφώς αναγνωρισμένα σαν ε, πιο ευαίσθητα, που έχουν ιστορικό βασανιστήριων, που είναι γυναίκες, παιδιά, συνόδευτοι ε, ανήλικες. Ε, όμως ε, ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ε, ιδιαίτερες ανάγκες στην αρχή. Μετά την κράτηση και λόγω των συνθήκων κράτησης γίνονται ευάλωτα άτομα και αποκτούν ειδικέ ανάγκες. Η κράτηση έχει απαξιωτικό αντίκτυπο στο, στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Κάνει τους ανθρώπους πιο αδύναμους και η ψυχική και πνευματική τους υγεία δεν δεν είναι πλέον τόσο καλή Βλέπουμε λοιπόν ότι ε, ένα άτομο είτε μπορεί να γίνει ευάλωτο, είτε η ευαλωτότητά του αυτή μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη, ξεκινώντας ακόμα και από την πρώτη εβδομάδα της ε, κράτησης. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι τα άτομα αυτά τα οποία ζουν σε κλειστά κέντρα, σε κέντρα κράτησης, μπορεί να παρουσιάσουν άγχος, συμπτώματα κατάθλιψης, μπορεί να έχουν ε, επίσης ε, κρίσεις οργής ή θλίψης, ε, λίθαργο, αισθήματα ενοχής, αισθήματα απόγνωσης. Υπάρχουν επίσης άλλες περιπτώσεις όπου λόγω της, των γλωσσικών φραγμών, λόγω της αίσθησης ότι δεν γίνεται κατανοητό το το πρόβλημα το άτομο αρχίζει να έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Ε, προβλήματα τα οποία διαρκούν ε, σε, στη μεγάλη πλειοψηφία 80 περίπου της 100 ακόμα και μετά την απελευθέρωσή τους. σε μερικές περιπτώσεις ο εγκλισμός ε, των ε, ε, ανθρώπων αυτών μπορεί να έχει μεγαλύτερη σκληρότητα όσον αφορά το, το πώς οι ίδιοι βλέπουν την κράτηση αυτή από ότι στους κρατούμενους του κοινού ποινικού δικαίου τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η μελέτη μας πραγματικά είναι ότι δεν θα πρέπει ε, τα άτομα αυτά να παραμένουν ε, σε κλειστά κέντρα και να κρατούνται. Ε, θα πρέπει να γίνονται ανεξάρτητοι έλεγχοι ήδη από την αρχή όσον αφορά τις ειδικέ ανάγκες ή τον ευάλωτο χαρακτήρα των ατόμων έτσι ώστε να μην υπάρξει κράτηση σε περίπτωση που το άτομο είναι ιδιαίτερα ευάλωτο. Ε, και έτσι ώστε να μην ε, γίνει ακόμα δυσχερέστερη η κατάσταση των ετούντων άσυλο. Βεβαίως, ε, επίσης να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, πληροφόρηση κατανοητή, καθώς επίσης και να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε δικαστική αρρωγή. Θα αναφερθώ τώρα σε εναλλακτικέ λύσει όσον αφορά ε, την κράτηση. Η μελέτη μας ε, καταδεικνύει ότι είναι πάντα αρνητικό θέμα η κράτηση. Ε, δεν αναφερόμαστε εδώ, δεν έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ένα κατάλογο ε, πρακτικών που μπορεί να είναι ορθές σε μία χώρα και λιγότερο ορθές σε μία άλλη. Ε, θεωρούμε ότι η κράτηση και οι συνθήκες κράτησης είναι ένα αρνητικό μέρος του, του συστήματος. Εμείς κάναμε την δική μας μελέτη, αλλά βασιστήκαμε και στα ευρήματα μιας οργάνωσης που λέγεται International Detention Coalition και που είναι μια οργάνωση ε, αυστραλιανή ε, και η οποία μετά από ε, μελέτη έχει προσπαθήσει να δει με ποιο τρόπο η κυβερνήσεις ε, μπορούν να βρουν εναλλακτικές λύσεις στην κράτηση, αν αυτές οι εναλλακτικές λύσεις κοστίζουν ε, περισσότερο και αν είναι πιο αποτελεσματικές και επίσης ε, πιο αντίκτυπο μπορεί να έχουν στα, στους ίδιους τους μετανάστες τα άτομα αυτά. συγγνώμη, οι εναλλακτικές λύσεις αυτές. τα σημαντικότερα βρήματα είναι ότι η δυνατότητα κράτησης αλλά χωρίς περιορισμό δηλαδή σε ανοιχτά κέντρα, ε, μπορεί να βελτιώσει πολύ την ε, κατάσταση. Ε, επίσης, λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλές μορφές αναλλακτικών λύσεων, η μελέτη καταδεικνύει ότι 80 με 90% των μεταναστών αισθάνονται πολύ καλύτερα σε αυτά τα ανοιχτά κέντρα. Κάποιες, ε, κάποια από τα καλύτερα τις ε, παραδείγματα μάλλον ε, βέλτιστης της πρακτικής είναι αυτά τα οποία αφορούν την κοινωνική αντιμετώπιση των των άσυλο και των μεταναστών. Στο Βέλγιο ας πούμε οι οικογένειες δεν κρατούνται πλέον αλλά μένουν σε κοινοτικά σπίτια και είναι συνδεδεμένες με έναν διαχειριστή της περίπτωσης τους που τους βοηθάει σε όλες τις διαδικασίες. Ε, επίσης ε, θεωρούμε ότι αυτές οι μελέτες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, έτσι, και να τις λάβουν τα κράτη υπόψη τους στην πολιτική ασύλου που ακολουθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τη συντομία σας. Έχουμε χρόνο για δύο-τρεις ερωτήσεις μονάχα, όχι παραπάνω. Γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσει και η διερμηνία. Κάποιο ερώτημα, ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι σίγουρος, σίγουρη ποιος από το πάνελ πρέπει να απαντήσει το ερώτημά μου. Κάποιος θα ήθελε ίσως να δώσει μια ε, απάντηση. Ναι. Ποια είναι η κατάσταση των προσφύγων ή των παράνομων μεταναστών που είναι υπό απέλαση, που προσπαθεί κανείς να, ε, ε, έχει κανείς την πρόθεση να τους απελάσει και οι οποίοι τίθενται σε ένα κέντρο κράτησης με κα, κανονικούς καταδίκους του ποινικού δικαίου. Υπάρχει ε, αυτή η πρακτική να αναμειγνύονται η προσαπέλαση μετανάστες με ποινικού καταδίκους ή όχι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ να σας πω συνολικά τι γίνεται, αλλά η εμπειρία μας είναι ότι υπάρχουν πραγματικά κέντρα κράτηση όπου γίνεται αυτή η ανάμειξη με κρατουμένους του κοινού ποινικού δικαίου. Πάρα, πολλοί, πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν αυτούς τους παράνομους, αν είναι παράνομοι μετανάστες, ότι είναι πραγματικά, ότι είναι, ε, ότι είναι σαν εγκληματίες γιατί έχουν παραβιάσει τον νόμο της χώρας μπαίνοντας παράνομα εκεί. Μπορώ να κάνω και μια συμπληρωματική. Έρχομαι από τις κάτω χώρες και η χώρα μου προσπαθεί να ποινικοποιήσει την παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα μου, αλλά δεν είχα κατανοήσει ότι υπάρχει η κράτηση αυτών των παρανόμων μεταναστών μαζί με καταδίκους. Είναι κάτι για το οποίο λοιπόν θα πρέπει να προειδοποιηθούν οι αρχές και άτομα όπως εγώ. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση στο Βέλγιο, λέει η κυρία Άκερ Αλλά εγώ θα ήθελα να σας προειδοποιήσω ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα συγκεκριμένα, δυστυχώς. Δεν μπορώ να σας δώσω πιο συγκεκριμένο. Κύριος Παπα-Νικολάου. Σύντομα ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε κέντρα κράτηση σε πολλές χώρες που δεν αντιμετωπίζουν με το κατάλληλο τρόπο τους, ε, τους κρατουμένους εκεί. Το ερώτημα είναι εκεί. Έχουμε και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να βελτιωθεί η κατάσταση στα κέντρα κράτησης. Θα μπορούσε να μου δώσει κάποιος μια απάντηση για το πόσο καλά δαπανώνται αυτά τα χρήματα, αν είμαστε αποτελεσματικοί στη χρηματοδότηση αυτή, αν υπάρχουν κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση της χρησιμοποίησης αυτών των κονδυλίων. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Δεν ξέρω για ειδικέ προτάσεις βελτίωσης των κέντρων κράτησης, αλλά σίγουρα οι καταστάσεις πάντα βελτιώνονται αν έχετε καλύτερη υποδομή. Σίγουρα υπάρχουν στην Ευρώπη περιπτώσεις κρατήσεως σε σοφρονιστικά καταστήματα. Στην Ιρλανδία το είδα αυτό, γυναίκες οι οποίες κρατούνται βρίσκονται κοντά σε δολοφόνους. Αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και πρέπει να αποφευθεί με κάποιο τρόπο. Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κράτησης, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε, σε, σε ανοιχτούς χώρους, σε χώρους αναψυχής, σε πληροφόρηση. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία βοηθούν να σπάσει η απομόνωση του χώρου κράτηση, αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο για να βελτιώσει κανεί τι συνθήκε και σίγουρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά, αλλά τελικά όλα αυτά είναι πολύ πιο πολυδάπανα από εναλλακτικέ λύσει που τα άτομα αυτά ενσωματώνονται σε κοινότητες, σε, ανοιχτούς, σε ανοιχτές συνθήκες. Είναι όλα αυτά πολύ καλύτερα γιατί τα κέντρα κράτης ακόμη και με τις βέλτιστες συνθήκες είναι σαν φυλακές. Ε, δεν θέλω να παραγνωριστεί μια παρέμβαση που έκανε προηγουμένως ο Βέλγος δικαστής, ο οποίος αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλάμε πολλές φορές για καταστάσεις οι οποίες είναι κοινωνικά και πολιτικά ακραίου χαρακτήρα. Και γι' αυτό δεν βλέπουμε το σύνολο του προβλήματος και η κοινωνία πολλές φορές δεν κατανοεί το σύνολο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων που έχει να κάνει με τα άτομα αυτά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να κάνουμε την προσπάθεια για να εφαρμόσετε στην πραγματικότητα τα δικαιώματα των ατόμων αυτών. Και ένα από αυτά τα οποία δεν ισχύουν είναι το δικαίωμα να υπάρχουν δύο επίπεδα ανέρεσης. Γιατί μιλάμε για τη διοικητική ε, απόφαση σαν πρώτο επίπεδο και την δικαστική σαν δεύτερο επίπεδο. Όχι, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο δικαστικά επίπεδα και πρέπει να υπάρξει και μία ενιαία αντιμετώπιση για τα θέματα αυτά. Όπως είπε ο Βέλγος ε, δικαστή δεν μπορεί να έχουν 30 δικαστέ 30 διαφορετικέ νομολογίε. Θα πρέπει να υπάρξει μια ενοποίηση στην ομολογία και όλα αυτά πρέπει κάποια μέρα να γίνουν ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αγωνιστεί να ενσωματωθούν σε μελλοντικά νομοθετήματα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Ρουι Ταβάρες, ο οποίος θα πρέπει να αναλάβει το επόμενο πάνελ, γιατί και το δικό του θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θα ήθελα να του φάω το χρόνο. Ρουί, έχει το λόγο και την Προεδρία. la montre. Le, le, le, le programme. Non. Ah, la montre, oui.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 Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Ω εισηγητή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το κοινό πρόγραμμα επανεγκατάσταση Ευρωπαϊκή Ένωση και τη τροποποίηση του Ευρωπαϊκό Ταμείου Προσφύγων, με χαρά ε, αναλαμβάνω να συντονίσω τη συζήτηση για τα θέματα αυτά. Ιδίω δε τη συγκεκριμένη στιγμή τη διαδικασία συναπόφαση η διαδικασία συναπόφασης ε, ως ε, γνωστόν ε, καθυστέρησε περισσότερο από όσο περιμέναμε. Το 2010, το Μάιο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τις δύο αυτές τις εκθέσεις με πολύ μεγάλη πλειοψηφία Υπήρξε συνεργασία μεταξύ των πολιτικών ομάδων και εγώ ως εισηγητής ε, συνεργάστηκα με τους κοιόδης ε, εισηγητές. Ε, υπήρχε μία έκθεση για την τροποποίηση, της τροποποίησεις στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας που δεν θεωρήσαμε ότι είναι τόσο κατεπίγουσα, αλλά παρουσίαζε ε, τις σκέψεις μας για ένα μελλοντικό πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Και εκεί ζητούσαμε μία ε, πραγματική υλοποίηση ενός προγράμματος επανεγκατάστασης Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητούσαμε αποτελεσματικότητα, ε, γρήγορη απάντηση στα θέματα επανεγκατάστασης και μας ενδιέφερε ιδιαίτερα να υπάρχει ένα μόνιμο τμήμα επανεγκατάστασης ε, κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του προγράμματος επανεγκατάστασης Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσε να διεξάγει βασικές αρμοδιότητες προτεραιότητας και να ε, βοηθά τα κράτη-μέλη και να παρακολουθεί στη συνέχεια την κατάσταση ώστε να έχουμε μεγαλύτερη ποιότητα στη διαδικασία της ε, ένταξης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Όλα αυτά τα περιείχε η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Η διαδικασία συναπόφασης μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Συνομοθετών, μας οδήγησε σε ε, αλληλεπικάλυψη των χρονικών ε, προγραμμάτων. Είχαμε το, ε, την βασική έκθεση για τις τροποποίησεις στο Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Προσφύγων και την έκθεση της πρωτοβουλίας και ξέρετε ότι δεν έχει περατωθεί ακόμα η διαδικασία. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες οι πολιτικές ομάδες ε, κατέληξαν σε κάποια συμφωνία επί του θέματος και υπήρχε και μεγάλη συνένεση στο Συμβούλιο ως προς τα βασικά ε, μέτρα ε, στα θέματα συναπόφασης. Επιπλέον κονδύλια σε θέματα επανεγκατάστασης για τα κράτη-μέλη, μια διπλή διαδικασία όπου θα υπήρχε ανακατηγορία, δηλαδή ανθρωπιστικές προτεραιότητες για τους περισσότερους ε, ε, πρόσφυγες, αλλά και αναπεριφέρεια, ε, όπου θα επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένες περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες θα επιλόγουμε και από τις αξιολογήσεις του Ταμείου Προσφύγων και των άλλων υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα προσφύγων. Δυστυχώς από το Μάιο του 2010 για θεσμικούς λόγους έχουν σταματήσει τα πράγματα και έχει ήδη χαθεί ένας χρόνος σε θέματα επανεγκατάστασης και μάλιστα στις παρούσες συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό φυσικά είναι εις βάρος των ανθρώπων που βρίσκονται σε καταβλισμούς προσφύγων και για μας ε, ήδη από το 2010 ήταν πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε γιατί σταματούσαν όλες αυτές οι κατεπίγουσες ανάγκες λόγω του άρθρου 290 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γιατί υπήρχε το πρόβλημα με τις πράξεις κατεξουσιοδότηση. Επιτέλους βρήκαμε μια λύση στο θέμα των πράξεων κατεξουσιοδότηση και έχουν ξαναξεκινήσει οι διαδικασίες με το Συμβούλιο και ελπίζουμε να έχουμε μια συνέχεια σύντομα θα έχουμε μια νέα μορφή συναπόφαση με αντιπρόταση πλέον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δούμε ποιε είναι οι περιοχέ προτεραιότητα χωρί να έχουμε και πράξει κατά εξουσιοδότηση. Εμείς λοιπόν ω εισηγητέ και σκιώδη εισηγητέ, απαντήσαμε πολύ γρήγορα στο Συμβούλιο στην όλη αυτή διαδικασία στη διάρκεια των δύο ετών και γνωρίζω ότι όλοι θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να υπερκεραστούν αυτά τα προβλήματα μέχρι το Δεκέμβριο. Αλλιώ θα χάσουμε άλλη μια χρονιά στα θέματα επανεγκατάσταση που σημαίνει ότι μέχρι το 2010 ε, κανένας από τους πρόσφυγες βάσει των κατηγοριών που έχουμε καθορίσει δεν θα μπορούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα χαίρουν τις επιπλέον χρηματοδότησης ε, και γενικώ θα χαθεί όλη αυτή η όθηση που θα είχε δημιουργήσει η υπεράτωση της διαδικασίας συναπόφασης. Θα ήθελα λοιπόν να ε, χαιρετήσω τους ε, ομιλητές που έχουμε εδώ στο πάνελ, να σας παρουσιάσω. Έχουμε τον κύριο Ιωάννης Βανχεμούντ που είναι αρμόδιος για την πολιτική επανεγκατάσταση της ΥΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών ε, ασχολείται και με τις δυνατότητες επανεγκατάστασης και τη βελτίωση της ποιότητας και της ένταξης των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνούμε φυσικά όλοι ότι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εγκατάστασης σίγουρα θα βοηθήσει το έργο της ΥΠΑ της εδώ στην ε, Ευρώπη και ο Γιωχάνες Βαγκεμούντ ε, συνεργάζεται μαζί μας και σε όλο σκεπτικό και στο συντονισμό της διαδικασίας. Στη συνέχεια έχουμε τον κύριο Χόβιγκ Ετιαμεζιάν από την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών στην Τινησία. Ε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι αυτό το κοινό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τις δράσεις μας και θα δούμε και κάποιες εικόνες και κάποιες εμπειρίες ε, του κυρίου Ετιεμεζιάν στην Τουνησία Στη συνέχεια, εδώ εξ αριστερέν μου, έχουμε τον κύριο Γιάκοπ Νταμ από την Υπηρεσία Μετανάστευσης της Δανίας, ε, στο δεύτερο τμήμα προϊστάμενος και είναι και εδώ στη μονίμη αντιπροσωπεία της Δανίας στο Συμβούλιο. Όλοι ελπίζουν ότι η Δανία θα συνεισφέρει ε, στην ε, διαδικασία συναπόφασης. Γνωρίζουμε βέβαια ότι η Ιδανική Προεδρία θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει και ε, μαζί με την Πολωνική Προεδρία η Τριάδα των Προεδριών βοηθά και φυσικά θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα σε θέματα επανεγκατάστασης. Κατόπιν έχουμε την κυρία Μπάρμπαρα Τόμας, υπεύθυνη για τη μεταναστατική η πολιτική και τα θέματα που αφορούν τους πρόσφυγες, αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζει πάρα πολλά και έχει συνεργαστεί μαζί μας εδώ και αρκετό καιρό. Γνωρίζουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι η χώρα που επανεγκαθιστά τους περισσότερους πρόσφυγες κάθε χρόνο. τα 10 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, είναι υπεύθυνα για την επεκατάσταση, επανεκατάσταση 4.000 περίπου ατόμων ετησίως. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η βοήθεια και οι ε, συμβουλές των ΗΠΑ θα είναι χρήσιμα. Και τέλος έχουμε τον κύριο Τόρστεν Μόριτς από την Επιτροπή των Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη, εκτελεστικός γραμματέας για την πολιτική και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εργάζεται εκεί από το 2002. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση λοιπόν να ξεκινήσει η συζήτηση, να δώσουμε το λόγο λοιπόν στον κύριο Φάνχεμουντ καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία παρουσίαση PowerPoint, αλλά ε, ίσως ε, είσαστε ήδη κουρασμένοι. Θα προσπαθήσω να προχωρήσω σχετικά γρήγορα. Έχουμε δύο επίγουσες εκκλήσεις να κάνουμε, μία προς τα Ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία προς τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτού κάνω αυτή τη διπλή έκκληση όμως, την κατεπίγουσα αυτή έκκληση, θέλω να κάνω ένα βήμα προς τα πίσω και να σας ε, εξηγήσω το πλαίσιο της επανεγκατάστασης και το γιατί η επανεγκατάσταση είναι τόσο σημαντική και πράγματι απαράγραπτη στο έργο του, της ε, αρμοστίας για τους πρόσφυγες. Θέλουμε να δώσουμε προστασία σε 10,5 εκατομμύρια πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο. 80% αυτών των πρόσφυγων ζουν σε φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες και αυτό είναι σημαντικό να το ξέρουμε. Πάνω από 8 εκατομμύρια λοιπόν βρίσκονται σε πολύ φτωχές αναπτυσσόμενες χώρες. Προσπαθούμε να έχουμε μόνιμες λύσεις για τα άτομα αυτά που θα τους δώσουμε. Υπάρχουν τρεις κατευθύνσεις που ακολουθεί η πατιαρμοστία. Για κάποιους κάποτε θα υπάρξει η εθελοντική, ο εθελοντικός επαναπατρισμός τους θα μπορούσαν να γυρίσουν στις αιστείες τους με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Για κάποιους άλλους τοπική ενσωμάτωση στη χώρα που τους παρέχει άσυλο. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν έχουν ζήσει γενιές στα στρατόπεδα προσφύγων και δημιουργείται μια δυνατότητα να ε, ενσωματωθούν. Αυτό δεν είναι τόσο συνηθισμένο όσο ο επαναπατρισμός. Η τρίτη λύση είναι η επανεγκατάσταση και πάλι είναι μια λύση που αφορά μονάχα λίγα άτομα, αλλά είναι μια σημαντική λύση. Και η δική μου πρακτική, εγώ έχω εργαστεί στην Ιεμένη ε, που είναι μια από τις τόσο φτωχές αυτές αναπτυσσόμενες χώρες, 152η σε δίκτυα ανθρώπινης ανάπτυξης μεταξύ 170 χωρών και αυτό είναι εύγλωτο ήδη. Η ΕΜΕΝ ήταν η μόνη χώρα που υπέγραψε την σύμβαση της Γενέβης από, την, ε, από τον αραβικό χώρο και είχε ανοιχτή πολιτική εναντί της Σομαλίας και των Σομαλών προσφύγων από την άλλη πλευρά του κόλπου του Άντεν. Ήταν λοιπόν ένα περιβάλλον που έδωσε στους πρόσφυγες δυνατότητα να ζουν είτε σε καταβλισμούς είτε σε αστικές περιοχές. Αλλά υπήρξε πράγματι η απόφαση της κυβέρνησης να δώσει προστασία σε αυτούς τους πρόσφυγες από τη Σομαλία αλλά και από την Αιθιοπία την προστασία του πρόσφυγα. Και εμείς προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για πολλούς όμως από αυτούς τους Σομαλούς, ε, Αιθίωπες ή Ερυθραίους, δεν υπήρχε δυνατότητα να επανέλθουν στη χώρα τους, ούτε καμιά δυνατότητα για τοπική ενσωμάτωση. Επομένως η επανεγκατάσταση ήταν και εξακολουθεί να είναι μια σημαντική λύση για τους πρόσφυγες στην Ιεμένη. <coughs> Δεν είναι μόνο μια λύση. Μπορεί να είναι και ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας. Όταν οι πρόσφυγες κινδυνεύουν να επαναπροωθηθούν στη χώρα προέλευσής τους όπου μπορεί να τύχουν εκεί καταδίωξης ή όταν η κατάσταση στη χώρα του ασύλου είναι τόσο επικίνδυνη που δεν μπορούν να μείνουν εκεί, τότε η επανεγκατάστασή τους είναι η λύση και ο τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η ασφαλειά τους. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η επανεγκατάσταση για τους, πρόσφυγε για τους πρόσφυγες αυτούς, αλλά όχι μόνο για αυτούς. Είναι σημαντική αυτή η δυνατότητα και για αυτούς οι οποίοι παραμένουν πίσω στις χώρες ασύλου. Μπορεί να έχει στρατηγικό αντίκτυπο. Μπορεί να ανοίξει πόρτες για αυτούς οι οποίοι ζητούν άσυλο και προσπαθούν να μπουν σε μια χώρα, εάν μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε στη χώρα που παρέχει άσυλο ότι δεν είσαστε μόνοι σας, η διεθνής κοινότητα σας βοηθάει για να βοηθήσετε αυτούς τους πρόσφυγες. Μπορεί να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, κάτι που δεν γίνεται συχνά, σας το λέω, αλλά προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό, μπορεί να είναι τμήμα μια συνολικής λύσης για όλους τους πρόσφυγες. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα στην Τανζανία όπου υπήρξαν πρόσφυγες από τον Μπουρούντι μετά τις τραχές του 1972 και έχουν ζήσει για γενιές στην Τανζανία. <clears throat> και τώρα λίγες χιλιάδες έχουν μπορέσει να επιστρέψουν σαν αποτέλεσμα μιας συνολικής λύσης και συμφωνίας των κυβερνήσεων. Κάποιοι από αυτούς μπόρεσαν να γυρίσουν στον Μπουρούντι. Κάποιοι έχουν επανεγκατασταθεί και πολλές χιλιάδες, ε, ελπίζουμε περίπου 70.000, θα πάρουν την υπηκότητα της Τανζανίας στα, στα επόμενα χρόνια. Αλλά αυτό σας δείχνει ότι η επανεγκατάσταση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για τους πρόσφυγες σαν τμήμα μιας συνολικής λύσης. Σαν τμήμα λοιπόν της καθημερινής μας εργασίας, αναζητούμε λύσεις για τους πρόσφυγες και κατά την ε, διακρύβωση της, του καθεστώτος τους και κατά τη διάρκεια της ε, παροχής συμβουλών βλέπουμε πολλές φορές ότι η επανεγκατάσταση μπορεί να είναι η μόνη λύση για κάποιους πρόσφυγες. Αυτή η διαδικασία ταυτοποίησης και αναγνώρισης συνεχίζεται και βλέπετε εδώ πέρα σε αυτό το βιβλίο που καλύπτει όλο τον κόσμο τα στοιχεία για όλες τις χώρες όπου υπάρχουν πρόσφυγες. Αυτό το βιβλίο, αυτή η έκδοση έγινε τον Ιούλιο και αναφέρει τις εκτιμόμενες ανάγκες επανεγκατάστασης σε όλες τις χώρες αυτές. Για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια προβλέπεται ένας αριθμός 780.000 προσφύγων, αλλά για του χρόνου, το 2012, οι αυτοί που πρέπει να έχουν προτεραιότητα για την επανεγκατάστασή τους είναι 172.000 στον αριθμό. Έχουμε λοιπόν τα 10,5 εκατομμύρια προσφύγων <clears throat> που είναι στην εντολή της ΥΠΑ της ε, αρμοστίας και 780.000 που θα χρειαστούν στα επόμενα χρόνια να επανεγκατασταθούν. Και τώρα να το συγκρίνουμε για με τον αριθμό των προσφύγων που επανεγκαθίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το 2010, 4.707 άτομα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αναφέρομαι τώρα στα προγράμματα ad hoc, και εκεί η Γερμανία επανεγκατέστησε ένα σημαντικό αριθμό προσφύγων πέραν αυτών που αναφέρονται εδώ. Η Γερμανία δεν έχει κάποιο πρόγραμμα εδώ στο, στην επανεγκατάσταση και επομένω δεν αναφέρεται εδώ, αλλά η ποσόστοση για το 2011 είναι 4.940, περίπου 5.000 από τις 780.000 που θα χρειαστούν επανεγκατάσταση. Αν το θέσουμε αυτό τώρα σε ένα γενικότερο πλαίσιο επανεγκατάστασης. Βλέπετε στο, με, το κόκκινο χρώμα τι κάνουν οι, όλες οι άλλες χώρες και με το μπλε, αν φαίνεται καθόλου, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι κολακευτικό αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι άλλες χώρες, 54.000 επανεγκαταστάθηκαν στις ΗΠΑ το 2010 που έχει ένα μέγιστο αριθμό 70 ή 80 χιλιάδες προσφύγων που μπορεί να επανεγκαταστήσει ένα χρόνο, αλλά 50-60 χιλιάδες είναι ρεαλιστικά νούμερα για τις ΗΠΑ, πολιτειες Πολιτείες, 6-7 χιλιάδες στον ε, Καναδά και ένας μικρότερος αριθμός στην Αυστραλία. συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει και αυτή κάποιο ρόλο και υπάρχουν χώρες με μακρά παράδοση όπως είναι η Σουηδία, η Δανία και η Φιλανδία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το εκτιμά ιδιαίτερα η πάτη αρμοστία για τους πρόσφυγες και μιλάει για συνολικούς έτοιμους. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι εδώ υπήρξε μια μικρή αύξηση το 2009 όχι μόνο στο κόκκινο αλλά και στο μπλε. Αυτό χάρη στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Νοέμβριο 2008 για να επανεγκατασταθούν 10.000 πρόσφυγες από το Ιράκ. Σχεδόν επετέχθη αυτό και αυτό δείχνει τη μεγάλη, της, το μεγάλο δυναμικό που υπάρχει. Υπήρξαν τα προγράμματα αυτά ad hoc και ιδίω η γερμανική κυβέρνηση δέχτηκε 2.500 πρόσφυγες μέσα σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Από το 2008 λοιπόν μπορούμε να πούμε <clears throat> ότι υπήρξε ένα σημείο καμπής και τα πράγματα έχουν αρχίσει να κινούνται. Υπήρξε μια αύξηση στην ε, ταχύτητα με την οποία γίνεται η επαναγκατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν νέες χώρες επανεγκατάστασης που μπαίνουν στην ε, παγκόσμια οικογένεια. Η Τσεχική Δημοκρατία, η Ρουμανία και η Ισπανία και η Βουλγαρία ανακοίνωσαν νέα προγράμματα το 2010. Θέλω να τονίσω λοιπόν ότι υπάρχουν εξελίξεις όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Μπορεί κανείς να δει μια αυξανόμενη αλληλεγγύη μεταξύ, μέσα στους δήμους, στις τοπικές ΜΚΟ, την κοινωνία των πολιτών, υποστηρίζοντας την επανεγκατάσταση και σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα να διαδραματίσουν ένα ρόλο για την υποδοχή των προσφύγων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό η διαδικασία <clears throat> επανεγκατάστασης δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς σωστή υποδοχή και χωρίς σωστή ενσωμάτωση. Και φυσικά σε τοπικό επίπεδο οι δήμοι, οι και οι τοπικές οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Στη Γερμανία υπήρξε μια πρόσφατη εκστρατεία, μια, ένα δίκτυο δήμων θέλουν έχουν οργανωθεί για να παίξουν ένα ρόλο στην επανεγκατάσταση και ασκούν πίεση στο ομόσπονδο κράτο για να παίξει πιο μεγάλο ρόλο σε αυτές τις ενέργειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί αυτές τις πρωτοβουλίες μέσω ενός ε, κοινού ε, ταμείου για τους, του Ταμείου για Πρόσφυγες και υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για το δίκτυο των Δήμων που ήταν μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Πάτη Αρμοστία είναι ευγνώμων προς το Κοινοβούλιο και προς τον εισηγητή του Κοινοβουλίου για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν στο θέμα αυτό. Λέγεται εδώ ότι αυτό χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, αλλά στην πραγματικότητα είναι πιλωτικό πρόγραμμα, οπότε έχει χωριστή χρηματοδότηση. Αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ για την ύπαρξη αυτού του πιλωτικού προγράμματο Ξαναγύριζω στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέφερε ο εισηγητής ήδη ότι υπάρχει μια θεσμική εμπλοκή σε σχέση με το κοινό πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρατάει ένα-δύο σχεδόν χρόνια αυτή η κατάσταση εμπλοκής και αυτό με ξαναφέρνει στην ε, κατεπίγουσα έκκλησή μου για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιτακτικό να υπάρξει μια λύση όχι σύντομα αλλά το ταχύτερο δυνατό. Και σας υπενθυμίζω <clears throat> την ε, ταινία Καζαμπλάνκα που είναι η πιο περίφημη ταινία για τους πρόσφυγες ότι χρειαζόμαστε μια λύση αν όχι σήμερα, αύριο ή μεθαύριο, μέχρι το Μάιο ή Ιούνιο του 2012, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτή είναι η στιγμή που οι χώρες οι οποίες δέχονται επανεγκατάσταση μπορούν να υποσχεθούν αριθμό προσφύγων για τη συνέχιση του παγκοσμίου προγράμματος. Αν λοιπόν οι χώρες αυτές δεν μπορούν μέσα στη νέα προσπάθεια η οποία ξεκινάει να υποσχεθούν θέσεις για επανεγκατάσταση και που δίνει τη δυνατότητα σε περαιτέρω χρηματοδότηση, τότε θα χαθεί αυτή η ευκαιρία. Δεν θα υπάρξει ένα πρόγραμμα το 2013 για να αντιμετωπίσει τα άτομα αυτά και τα πράγματα θα μείνουν μπλοκαρισμένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να μείνει πίσω από του άλλου. <clears throat> το πρόγραμμα αυτό μπορεί να είναι ωραίο, αλλά είναι ένα μικρό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα εθελοντικό, είναι ένα πρόγραμμα πλαίσιο. Ελπίζουμε ότι οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν τουλάχιστον αυτό το πρόγραμμα να το εφαρμόσουν στου επόμενους μήνες. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε περισσότερες θέσεις επαναγκατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ένα πιο έντονο ρόλο να παίξει για την επανεγκατάσταση και μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λύση αυτή πιο στρατηγικά. Υπάρχει προσθέμενη αξία λοιπόν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως όχι με τους τωρινούς αριθμούς, αλλά όταν υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός, τότε θα έχει επανεγκαθιστόμενο, θα έχει μεγαλύτερο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα κάτι άλλο, θέλω να ξεκινήσω για να πω κάτι τα οποία θα συνεχίσει ο συνάδελφός μου από την Τινησία Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σχετικά μικρό αριθμός προσφύγων στην Βόρεια Αφρική, περίπου 5.000 άτομα τα οποία χρειάζονται επανεγκατάσταση, αλλά πρέπει να είναι ταχεία και επίγουσα αυτή η επανεγκατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφερε 10.000 θέσεις για το Ιράκ, γιατί όχι 5.000 από τη Βόρεια Αφρική. Οι Ηνωμένε Πολιτείε προσφέρουν ένα ανοιχτό αριθμό ε, θέσεων, αλλά οι διαδικασίε στι ΗΠΑ είναι πάρα πολύ βραδίε. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καλύψει το κενό. Θέλω να σα ευχαριστήσω και σα δείχνω μια οικογένεια από το όρομο που ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2006 ως πρόσφυγες από την Αιθιοπία και μένουν τώρα στο Μπράιτον. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι παρίστανται ε, άτομα τα οποία έχουν διαφορετικό βαθμό έκθεσης ε, στο θέμα της επανεγκατάστασης. When he said that in a year the needs for settlement could be uh, Αυτά που μας είπε λοιπόν ο κύριος Βαν Χεμούντε ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για μας που έχουμε ασχοληθεί ε, με το θέμα της ε, πανεγκατάστασης, Ξέρουμε ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω από τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες. Είχαμε βέβαια και παλιότερα θέσει πολύ φιλόδοξους στόχους, ας πούμε στην ε, Σουηδική Προεδρία θυμάμαι ότι είχαμε πει ότι θα διπλασιάσουμε ε, τους αριθμούς, ότι θα έχουμε 5.000 ε, ανθρώπους σε επανεγκατάσταση κτλ. αλλά υπάρχουν ζητήματα τα οποία άπτονται του ασύλου, της επανεγκατάστασης που είναι εξαιρετικά ε, περίπλοκα. 200.000 μπορούμε να τις φτάσουμε εάν όλοι, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συντονισμένα ε, ασχοληθούν. Και αναφέρομαι εδώ στα Ηνωμένα Έθνη, στη Βενεζουέλα, στη Βραζιλία, ε, στην Χιλή κτλ. Πιστεύουμε ότι εάν έχουμε φιλόδοξους στόχους και αν συντονίσουμε τη δράση μας, μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Και ενδεχομένως και πριν τον Ιούνιο ακόμα, να καταφέρουμε να έχουμε ε, ήδη μία πρώτη συνάντηση των εμπειρογνωμόνων τον Ιανουάριο και μετά να έχουμε μέχρι τον Ιούνιο και την ε, ε, πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου σχετικά ε, με την οδηγία και σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής και επομένως μέχρι τον Ιούνιο να έχουμε ε, συγκεκριμένα ε, ζητήματα λύση. Εμείς θέλουμε μέχρι το τέλος του 2012 να έχουμε τελειώσει την ανάπτυξη της οδηγίας. Ευχαριστώ πολύ. Τον κύριο, δίνω τώρα το λόγο στον κύριο Τιεμεζιάνου. Ευχαριστώ πολύ. Πριν σας δείξω ε, κάποιες ε, φωτογραφίες, θα ήθελα να σας δώσω μια ιδέα για το τι εννοούμε όταν λέμε ότι οι καταστάσεις είναι επίγουσες. Οι ποινήσιοι έδωσαν σε όλους μας ένα παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο δούλευσαν σε μια χώρα που δεν έχει κυβέρνηση, ε, που δεν έχει κοινή στρατηγική, ε, που όμως ε, δούλεψε σε ανθρωπιστική βοήθεια και κατάφερε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του εκατομμυρίου αυτού που, των ανθρώπων που προσπαθούσαν να φύγουν από την Λιβύη, καθώς επίσης και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ταξιδιωτών ή μεταναστών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Ε, η αλληλεγγύη που εδείχθη απέναντι σε ε, υπηκόους 64 και πλέον ε, χωρών ήταν εξαιρετική. Χώρες που μέχρι τότε οι Τινήσοι περίπου δεν ήξεραν ότι υπάρχουν. Αυτές είναι πρώτες φωτογραφίες εκατοντάδων ανθρώπων που συνοθούνται στα σύνορα Λιβύης Τινησίας. Ε, φιλοξενήθηκαν σε νοσοκομεία, σε ε, σχολεία από τους τινήσιους αλλά ε, κάποια στιγμή δεν έφταναν πια ούτε αυτά τα κτίρια και έπρεπε να βρεθούν άλλες εναλλακτικές λύσεις. Επομένως, η αρμοστία και άλλοι ε, προσπάθησαν να βρουν λύσεις. Δημιουργήθηκε λοιπόν ε, ένα στρατόπεδο, ε, αρχικά στρατόπεδο μόνο μεταναστών και μετά και προσφύγων στο μέσο της ερήμου άνθρωποι από τελείω διαφορετικέ συνθήκε από πολλέ χώρε. Ήταν χειμώνα, παρόλα αυτά του βλέπετε, κάνουν μπάνιο έξω και ο συντονισμός έγινε όλος από την, την Ισία. και όλος ο εξοπλισμός και η ανθρωπιστική βοήθεια ε, έφτανε από την Τίνιδα. Βεβαίω έπρεπε να ξεκινήσει κάποια στιγμή και η διαδικασία επανεγκατάστασης, δηλαδή επιστροφής των ανθρώπων αυτών εις ε, την, ε, στις χώρες τους. Ε, κανείς βέβαια δεν ρώτησε την Τινησία εάν είχε την δυνατότητα να διώξει με οργανωμένο τρόπο αυτούς τους ανθρώπους και ε, αναγκάστηκαν λοιπόν να αυτοσχεδιάσουν άνθρωποι οι οποίοι ποτέ δεν είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με μια τέτοια ανθρωπιστική ε, επίγουσα κατάσταση. Αυτό είναι ένα άλλο μάθημα που ε, μάθαμε από τους της ε, Επίσης ε, ε, πρέπει να πούμε ότι ήταν ε, άνθρωποι οι οποίοι ήδη έφεραν τραύματα ψυχολογικά και άλλα από τις καταστάσεις που άφηναν τις εμπόλεμες χώρες κτλ. και που είχαν χάσει τα πάντα, ε, ζωές οικείων και ε, περιουσιακά στοιχεία και βρέθηκαν ε, σε αυτό το στρατόπεδο όπου έγιναν ακόμα μεγαλύτερες, έγινε ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημά τους. Άνθρωποι οι οποίοι βέβαια στα στρατόπεδα αυτά αισθάνονται ότι εξαρτώνται από τους άλλους προσπαθούν να βρουν ένα μηχανισμό αντίστασης ε, και καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκε διαβίωση στην έρημο ε, όξυναν ακόμα περισσότερο το πρόβλημά τους. Γι' αυτό λοιπόν, βλέποντας ότι υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να βοηθηθούν, ε, ξαναχτίσαμε, ξαναστήσαμε το στρατόποδο της Σούσα. Ε, και βεβαίω ε, η προφανής ερώτηση ήταν «Μα γιατί μας χαραβάζετε στο στρατόπεδο, γιατί δεν μπορείτε να μας επανεγκαταστήσετε ε, γρήγορα». Αναφέρομαι εδώ στο όχι στους μετανάστες που γύρισαν στα σπίτια τους. Μιλάμε για Σομαλούς, για Ερυθρέου, οι οποίοι δεν μπορούν να γυρίσουν στις χώρες τους, Λιβύους που δεν μπορούν να επιστρέψουν στη Λιβύη. Άρα μιλάμε για πρόσφυγε και αιτούντες άσυλο. Κοιτάξτε, μπορεί να προσπαθήσουμε να ξαναχτίσουμε και να ξαναστήσουμε το στρατόπεδο, αλλά ε, οι συνθήκε διαβίωση στην έρημο είναι πάρα πολύ δύσκολε. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι Λίβοι, α πούμε, ήταν ε, από αστικού πληθυσμού. Δεν ε, είχαν ζήσει όλη του τη ζωή σε πόλει. Δεν ήξεραν πώ να λύσουν, πώ να ζήσουν στην έρημο, πώ να ζήσουν έτσι και οι καταστάσεις που αντιμετωπίζουν είναι εξαιρετικά δύσκολες. Ε, προσδοκούμε λύση και ε, το εύχονται όχι μονάχα ε, όσοι διαμένουν στο στρατόπεδο, αλλά και οι τινήσιοι και οι τινησιακές αρχές. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πληθυσμό 4.000 ανθρώπων στο στρατόπεδο και στρέφονται όλοι προς εμάς και μας λένε «Μα τι κάνετε εσείς, τι κάνει η διεθνής κοινότητα γι' αυτό» Ε, σας δείχνω εδώ κάποιες φωτογραφίες ε, οι οποίες δείχνουν ότι προσπαθούν να βρουν μια ομαλότητα και μια ομαλή καθημερινότητα ε, όσοι ζουν σε αυτό το στρατόπεδο. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ηλεκτρισμός, πράγμα όχι συνηθισμένο για αυτά τα στρατόπεδα, αλλά και αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Και μάλιστα πριν από μια εβδομάδα είχαμε και πλημμύρες. Ε, μετά από καταρακτώδεις βροχές ε, αναγκαστήκαμε να ε, ξαναστήσουμε, να κλείσουμε παραπάνω από το μισό του στραθοπέδου και εκεί προκαλέσαμε περαιτέρω προβληματισμό στους κατοίκους. Επίσης εκεί είχαμε και ένα ευχάριστο νέο από την πλευρά της ε, Νορβηγίας, ένα πρόγραμμα νορβηγικό, βλέπετε, δείτε τις σχετικές εικόνες. Και βεβαίως μέχρι εσείς ως διεθνής κοινότης να αποφασίσετε ότι θα κάνετε κάτι, ε, αυτοί οι άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να περιμένουν. Βλέπετε εδώ ε, κάποιες χαρούμενες στιγμές. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ήμουν κοντά στους ε, πρόσφυγες από τον ε, Φεβρουάριο μέχρι τώρα και είναι συγκλονιστικό ας πούμε να βλέπεις έναν γιατρό από τη Σομαλία ο οποίος μετά από, τόσες, ε, από τόσους μήνες και τόσες τελεπορίες μπορεί να ελπίζει ότι θα ξαναχτίσει τη ζωή του σε μια άλλη χώρα. Θα ήθελα να θίξω και κάποια ζητήματα μαζί σας σήμερα. Ένα η κατάσταση στο στρατόπεδο ε, θα δυσχεράνει περαιτέρω γιατί ενσκύπτει χειμώνας. Δεύτερον, ότι οι αριθμοί δεν είναι πάρα πολύ μεγάλοι, επομένως από τεχνικής απόψεως μπορεί να βρεθεί κάποια ε, λύση ε, και επίσης εμείς είμαστε έτοιμοι όσον αφορά τις νομικές διαδικασίες. Η νομολογία τον Δεκέμβριο θα είναι έτοιμη. Επομένως δεν περιμένουμε από εσά κάποια κίνηση. Επίση, δεν είναι δυνατή σε αυτή την περίπτωση η ενσωμάτωση με τον τόπιο πληθυσμό. Ε, έχουμε ανθρώπου από την Ουγγάντα, από τη Σομαλία, από την Ερυθρέα που δεν μπορούν να βρουν την θέση του στην Τινησία. Δεν είναι δυνατόν, δεν πρόκειται να γίνει και επομένως ε, ευθύνη μας ε, και ευθύνη όλων ε, είναι να τίνουμε χειραβοηθείας προς τους την και να τους πούμε εσείς αναλάβατε να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες ενός εκατομμυρίου, μπορούμε να σας βοηθήσουμε για να καλύψετε τις ανάγκες τριών-τεσσάρων χιλιάδων. η διεθνή κοινότητα και οι ανθρωπιστικέ οργανώσει ε, εξακολουθούν ε, βεβαίω να βοηθούν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περίπου 700.000 Λίβοι ε, είχαν φιλοξενηθεί για κάποιο διάστημα στην Τινησία και εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα καμιά 25.000 οι οποίοι δεν μπορούν να ε, επιστρέψουν στην ε, ε, Λιβύη. Δηλαδή τώρα έχουμε το ανάποδο κάποιους, κάποιες χιλιάδες Λιβύων που λόγω της αντιστροφής, της ανατροπής ας πούμε του, του καθεστώτος του Καντάφη στην Λιβύη και της νέα, του νέου καθεστώτος δεν μπορούν πλέον να επιστρέψουν στην Λιβύη. Επομένως εξακολουθούμε να έχουμε στρατόπεδα για τους ανθρώπους αυτούς και, και κοστίζει πολύ. Ε, ε, επομένως θα πρέπει κανείς να κατανοήσει ποιο είναι το κόστος το οποίο έχουν αναλάβει οι τινήσιοι. Και συγκριτικά είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τελευταίο σημείο. Ενδεχομένως ε, υπάρχει ανάγκη να καταδειχθεί στους τινησίους ότι δεν ε, έκαναν λάθος ε, που έδειξαν αλληλεγγύη και υποδέχτηκαν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να τους πείσουμε ότι ε, έκαναν το σωστό. Ε, και επομένως ε, τώρα που πλησιάζει ο χειμώνας ε, το στρατόπεδο της Σούσα θα γίνει πάρα πολύ δύσκολο και επομένως εγώ τι να σας πω, εγώ μένω στο Ζαρζής, δεν το σπίτι μου, έχω σπίτι κανονικό, δεν μένω στη Σούσα, αλλά μην ξεχνούμε ότι χρειάζεται βοήθεια έτσι ώστε να φύγουν οι άνθρωποι από το στρατόπεδο της Σούσα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι εκπληκτικά τα όσα διαπιστώνουν αυτοί που έρχονται απ' έξω, δεν είναι εκεί στο στρατόπεδο της Όσα. Σε κάποια ε, στρατόπεδα ε, βλέπετε ότι έχουμε παιδιά και όταν τους ρωτήσουμε γιατί θέλουν να επανεκατασταθούν μας λένε ότι έχουμε χάσει τα πάντα αλλά το μόνο μας κεφάλαιο θα είναι παιδεία. Γι' αυτό ακριβώς και διοργανώνουμε μαθήματα για τα παιδιά. Ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο διαπίστωσα και από τις φωτογραφίες που είχατε ε, ε, να μας δείξετε τα καλά νέα για το ε, πρόγραμμα για την κατεπίγουσα επανεγκατάσταση που δεν είναι το ίδιο με το πρόγραμμα για τους Δήμους που ανέφερε ο κύριος Πανχεμούντ ε, έχει εγκριθεί εδώ και δύο εβδομάδες από την Επιτροπή Προϋπολογισμών και ε, θα εγκριθεί και από την Ολομέλεια και είναι επιπλέον 2 εκατομμύρια για επίγουσα επανεγκατάσταση τα οποία κονδύλια μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Αυτό για την εφαρμογή των κανόνων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων. Επίσης, κάτι το ε, οποίο υπάρχει επίσης στη συναπόφαση και εκρεμεί ως προς την απόφαση, είναι ε, στρατόπεδα προσφύγων τα οποία έχουν ε, επληχθεί από φυσικές καταστροφές. Όταν ξεκίνησε η συζήτηση δεν ήταν τόσο προφανές ε, ότι θα τα καταφέρουμε και κάποιοι μας είπαν να μην το θέσουμε ως προτεραιότητα. Αλλά όπως βλέπουμε ήδη από τις φωτογραφίες της Σούσα ήδη υπάρχουν ζημίες από φυσικές καταστροφές και υπάρχει στα χαρτιά, ελπίζω να το υλοποιήσουμε κιόλα. Ελπίζω να είμαστε πιο πειθαρχημένοι με το χρόνο και να τηρήσουμε λίγο καλύτερα τα χρονικά όρια. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μόριτς, λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας ευχαριστώ διότι για, σε μια κρόαση για το κοινό σύστημα ασύλου έχουμε συμπεριλάβει και την ε, κατάσταση. Αν βλέπαμε πώς είχε τα πράγματα πριν από πέντε χρόνια θα διαπιστώναμε ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Για όσους δεν μας γνωρίζετε είμαστε η οργάνωση Ομπρέλα για την Επιτροπή των Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη Έχουμε ορθόδοξες, προτεσταντικές και αγγλικανικές εκκλησίες κυρίως που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πρόγραμμα επανεγκατάστασης και να πω ότι είμαστε υπέρ των αναγκών προστασίας ανεξάρτητα από τις εθνικές ε, ή θρησκευτικές καταβολές κάποιου. Η επανεγκατάσταση, όπως είπαν ε, ε, κάποιοι, είναι ε, λίγο ακαθόδε ζήτημα. Ε, υπάρχει ελάχιστη αν όχι και καμία νομική βάση ε, για το θέμα αυτό και αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αλλά και πολύ ενδιαφέρον γιατί το μόνο που έχουμε είναι η ισχύ των επιχειρημάτων μα και νομίζω ότι αυτό κατέδειξαν και τα όσα είπαν οι προλαλήσαντε προηγουμένω αν δούμε τις φωτογραφίες, αν έχουμε μεταβεί επιτόπου σε περιοχές όπως στο στρατόπεδο Σούσα ή σε άλλες περιοχές, είναι σαφές ότι απαιτείται η επανεγκατάσταση και παρόλα αυτά θα είναι, δεν θα είναι παρά μόνο σταγόνα στον ωκεανό. Θα πρέπει λοιπόν σαφώς να επισημάνουμε γιατί είναι απαραίτητη η επανεγκατάσταση στον κόσμο που ζούμε τη σήμερα ημέρα. ο πρόεδρο, ο οποίο ήταν εισηγητή για τα θέματα επανεγκατάσταση, άρχισε εξηγώντα όλες τις δυσκολίες. Και πολλές φορές εδώ ε, συχνά υπάρχει αίθηση έχει σταματήσει το θέμα, είναι πολύ δύσκολο, υπάρχει θεσμικό πρόβλημα. Ε, να σας πω όμως ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε και νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε ανεξάρτητα από το κατά πόσο θα προχωρήσει το ζήτημα που έχουμε στη συναπόφαση. Και έχω διάφορες εκθέσεις για το θέμα και υπάρχει μια εξαιρετική το ψήφισμα της 8 η Μαΐου του 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κοινό πρόγραμμα επαναγκατάστασης. Πολύ χρήσιμο το έγγραφο αυτό και εδώ υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μας ενθαρρύνουν όλους να συνεχίσουμε με αυτά που μπορούμε να υλοποιήσουμε. Καταρχάς υπάρχει το γεγονός ότι πολλά πράγματα είναι ε, ε, υπατμών αλλά χρειάζονται μια κάποια όθηση. Πρέπει να γίνει μια συζήτηση επί της πολιτικής, πρέπει να παρουσιαστούν και τα επιχειρήματα τώρα που τα χρειαζόμαστε. Και νομίζω ότι ένα από τα βασικά σημεία για μένα είναι το γεγονός ότι πρέπει να είμαστε τολμηροί και να λέμε πόσους ανθρώπους θα μπορούσε ε, να επανακαταστήσει σε ένα πλαίσιο 5-10 ετών. Ωραίο να λέμε για προτεραιότητες, αλλά αφού ε, μιλάμε για 5.000 ή 10.000 ε, ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι μόνο περιφερειακό ποσοστό. Υπάρχει νόημα για την επανεκατάσταση αν έχουμε οικονομίες κλίμακες, αν υπάρχει ένα ε, πρόγραμμα ε, πολύ μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Παραδείγματο Φάρη αναφέρεται συνέχεια ο αριθμός των 40.000 στις ΗΠΑ και καλό θα ήταν να επικεντρωνόμαστε σε αυτά και όχι στους αριθμούς που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και τότε έχει νόμιμα η επανεγκατάσταση. Πράγματι μπορούμε να μιλήσουμε τότε σε χώρες όπως η Τινησία και να τους πούμε ότι ε, έχουμε αποτελέσματα για σας. Αλλιώς λόγια στον αέρα λέμε και λυπάμαι που σας το λέω έτσι. Ε, συζητήθηκαν πολύ σημαντικά θέματα, ε, η χρήση κοινών υποδομών, ε, κοινή αξιολόγηση επανεκατάστασης που έχουμε να εξελίξει. Υπήρχε μια κοινή δράση, την πρωτοβουλία για το Ιράκ και εδώ θα ήθελα να πω ότι επειδή αυτό ήταν πιλωτικό πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μήπως θα έπρεπε τώρα να ξεκινήσει ένα νέο πιλωτικό πρόγραμμα και να απαντήσουμε στην κρίση που έχουμε στο κατόφλι μας, αυτή που αναφέρθηκε τώρα, στη Βόρεια Αφρική, δεδομένου ότι είναι μια πάρα πολύ περιορισμένη κλίμακα επιχείρηση και πραγματικά είναι στην πόρτα μας ε, και μπορεί να γίνει με πολλή βοήθεια από τις τοπικές κοινωνίες ε, στους ανθρώπους που θα λάβουν συνδρομή απευθείας εκεί αναφέρθηκαν οι συμπράξει σε δημοσίου και ιδιωτικό τομέα και διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν κάποια καλά παραδείγματα και σε τοπικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό πρέπει να φτάσει και στα κράτη-μέλη. Ανάπτυξη δομών συνεργασία ε, μεταξύ ιδιωτικού και δημότιου τομέα, τη ΥΠΑ τη Αρμοστία για, του ε, πρόσφυγε και τη κοινωνία των πολιτών. Γιατί σύντομα η κοινωνία των πολιτών θα διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο ε, ως ε, ε οι άνθρωποι που θα υποδέχονται τους ε, ανθρώπους που εγκαθίσταται. Και επίσης επισημαίνεται ιδιαίτερα η ανάγκη να υπάρχει ένα εξειδικευμένο τμήμα. Ε, κάποιοι λένε γιατί να το χρειαστούμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ε, βιώνουμε μια στρατηγική σημασία ε, χρονική συγκυρία. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν εδώ, αλλά από τις συζητήσεις που έκανα εγώ με τον κύριο Φύς και άλλους, δεν έχω κλάβει το μήνυμα ότι πρόκειται για μία ε, βασική προτεραιότητα, διακαή επιθυμία για το ε, προχωρήσει στο θέμα της ΕΑΣΟ. Κα... Τι, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της πολιτικής μας από την αρχή ο οργανισμός αυτός. Αναφερθήκαμε σε ευέλικτες προτεραιότητες, σε ξεκαθορισμό προτεραιοτήτων, ε, χώρες προσφύγων που θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα και εδώ νομίζω ότι αναφερόμαστε πάρα πολύ ε, στα τεχνικά στοιχεία ενός προγράμματος, πώς θα είναι η υποδοχή σε τοπικό επίπεδο, ε, αλλά το θέμα είναι γιατί υπάρχουν ομάδε που χρειάζονται προστασία, γιατί υπάρχουν ομάδε που χρειάζονται επανεγκατάσταση και σε ποιε ομάδε ανθρώπων αναφερόμαστε επακριβώ, διότι ορισμένε φορέ έχουμε μια πολύ μικρή ομάδα που αποτελεί προτεραιότητα για την επανεγκατάσταση, ώστε να μπορέσουν να υποφαληθούν και κάποιοι από την τοπική του ένταξη και από, την, από τον επαναπατρισμό του. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε κάποια πράγματα παραπάνω για την επανεγκατάσταση και εδώ τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση με πρώτο το Κοινοβούλιο μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Πολλοί αναφέρθηκαν και στην ομάδα πυρογνωμόνων για την επανεγκατάσταση. Είχαμε φανταστεί ότι αυτή η ομάδα θα διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο για τον καθορισμό προτεραιοτήτων. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο το ζήτημα αυτό, αλλά πολλά μπορεί να γίνουν από την ομάδα πυρογνωμόνων παρά το γεγονός ότι δεν χρειάζεται να μιλάμε μόνο για τις προτεραιότητες σε οικονομικό επίπεδο. Πολλέ από τις χώρες που ξεκίνησαν την επανεγκατάσταση την ξεκίνησαν γιατί είχαν την εμπειρία από άλλες χώρες, γιατί υπήρχαν γνώσεις, γνώριζαν ότι υπήρχε εμπειρογνωμοσύνη και μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν. Μία ομάδα λοιπόν εμπειρογνωμόνων, ακόμα και αν δεν αναφέρεται καθόλου στο οικονομικό το, ε, κομμάτι, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και είναι χρήσιμο. Σας αφήνω λοιπόν με αυτά και να σας πω ότι δεν θα πρέπει να κοιτάμε τι δεν μπορούμε να ελοπίσουμε και τι είναι πολύ δύσκολο, αλλά να δούμε τι μπορούμε να προωθήσουμε και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προλιάνει πολύ καλά το έδαφος και ελπίζω να το συνεχίσει αυτό το έργο και στην θεσμική συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Μόριτς. Θυμάμαι πολύ καλά αυτή την έκθεση. Γι' αυτό Αναφέρθηκα στην έκθεση πρωτοβουλία. Και θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Μασίπη Ντάλγο, την κυρία Χίρ, τη Σκακέλα από του Πράσινους, τον Γιώργο Παπανικόλα από το ΕΛΚ και κύριο Τίπκοφ από το συντηρητική ομάδα. Συνεργαστήκαν πολύ καλά σε αυτήν την ομάδα. Και κάτι περιλαμβάνει αυτή η έκθεση είναι η μονάδα επανεγκατάστασης στα πλαίσια του ΕΑΣΟ. Γιατί έχουμε τα χρήματα, δεν έχουμε τους απαραίτητους ανθρώπινους πόρους και δεν έχουμε και την ανθρώπινη αίσθηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν ε, θα έχουμε μια προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν για την επανεγκατάσταση στα πλαίσια της Ολομέλης και ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλά νέα από το Συμβούλιο στη συζήτηση αυτή. Αλλιώς θα πρέπει να συνεχίσουμε την πίεσή μας. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Τόμας από την ε, αποστολή των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως αναφέρθηκε, εγώ είμαι η αρμόδια στην ε, αποστολή της Ευρωπα... της... των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα μετανάστευσης και προσφύγων. Έχω σταθεί σε αυτή την θέση για τα τελευταία δύο χρόνια περίπου και στα πλαίσια της συνεργασίας μου με, την... με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κοινωνία των πολιτών έχω δει να υπάρχουν κάποιες σημαντικές διαφορές σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την επανεγκατάσταση. Και θέλω να σταθώ σε τρεις από αυτές τις πτυχές σήμερα. Ένα ενδιαφέρον σημείο για μένα είναι καταρχήν η συχνότητα με την οποία τα κράτη-μέλη <clears throat> θέτουν τη βασική ε, ευθύνη για την εγκατάσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών τους. Εγώ πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό οι... επηρεάζονται οι συζητήσεις και η συνέχεια που δίνεται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή το Υπουργείο για την εσωτερική ασφάλεια, Homeland Security, παίζει ένα σημαντικό ρόλο για την επιλογή και τον έλεγχο ασφάλειας για τους ε, πρόσφυγες οι οποίοι θα επανεγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θεωρείται ότι είναι κάτι το οποίο αφορά τόσο την εξωτερική μας πολιτική όσο και τις εσωτερικές μας πολιτικές. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Γραφείο για τους πρόσφυγες στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι αυτό το οποίο διατυπώνει την πολιτική μας σε σχέση με, το, με τους πρόσφυγες και συνεργάζεται και με άλλες υπηρεσίες μέσα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ ώστε οι, τα προγράμματά μας να ικανοποιούν και τους ανθρωπιστικούς στόχους μας και τους στόχους μας εξωτερικής πολιτικής. Όπως ακούσαμε σήμερα, οι, τα προγράμματα αυτά μπορούν να ανακουφίσουν την πίεση στις χώρες οι οποίες υποδέχονται πρόσφυγες και μπορεί να τους δώσει τη δυνατότητα να προσφέρουν άσυλο σε άλλους πρόσφυγες. Η επανεγκατάσταση μπορεί επίσης να βοηθήσει άλλες ανθρωπιστικές λύσεις, είτε είναι η πρόθεση της, ε, ε της, ε, <clears throat> του επαναπατρισμού τους ή της ε, τοπικής τους ενσωμάτωσης. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό από μία έποψη εξωτερικής πολιτικής είναι ότι όλα αυτά μπορεί να επηρεάσουν ευρύτερους στόχους εξωτερικής πολιτικής όπως είναι η ειρήνη και η σταθερότητα σε περιοχές σύγκρουσης. Η επανεγκατάσταση των προσφύγων δείχνει και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ στα ανθρωπιστικά θέματα, κάτι το οποίο μπορούμε, προσπαθούμε να το δείξουμε σαν παράδειγμα σε άλλους. Μια άλλη προσέγγιση των ΗΠΑ που διαφέρει από αυτά που έχω δει σε κάποιες άλλες χώρες είναι ότι χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα τις εταιρικέ σχέσεις κάτι που ανέφερε προηγουμένω ο Το πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών για την επανεγκατάσταση δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς τη συμμετοχή πολλών άλλων εταίρων σε διάφορα επίπεδα, εθνικό, τοπικό επίπεδο, ομάδες της κοινωνίας της πολιτείας, θρησκευτικέ ομάδες κτλ. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο εμπλέκεται το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, το, οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την εργασία, με τη στέγαση και με την παιδεία. Και ορισμένε από αυτέ τι υπηρεσίε έχουν ειδικά προγράμματα για του πρόσφυγε, αλλά συμπεριλαμβάνουν του πρόσφυγε σε γενικότερα προβλήματα που έχουν να κάνουν με του μετανάστε ή τι μειονότητε. ή ε, δίνουν έμφαση στην δυνατότητα των προσφύγων να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίε. Υπήρχε, υπάρχουν επίσης συμβόλαια με εννέα μη κυβερνητικέ οργανώσεις, 7 από τις οποίες έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα, για να βοηθήσουν την επανεγκατάσταση των προσφύγων. Όλοι αυτοί οι φορείς χρησιμοποιούν τα εσωτερικά τους δίκτυα σε εσωτερικό επίπεδο, παραγωγός χάρη η συνέλευση των καθολικών επισκόπων που μπορεί να λειτουργήσει μέσα από τα τοπικά της δίκτυα, η οργάνωση λουθυρανών ιερέων επίσης, και υπάρχει και η Διεθνής Επιτροπή για τις πρόσφυγες μέσω των τοπικών γραφείων τους. Όλες αυτές οι οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο μπορούν να βασιστούν στους, ε, στα μέλη τους σε τοπικό επίπεδο για βοήθεια. Πρόκειται για θρησκευτικέ ε, για ενορίες, για θρησκευτικέ οργανώσεις, για άτομα από κάθε προέλευση και κάθε επάγγελμα και επίσης συμμετέχουν στο να κάνουν ράνους για να μπορέσουν να συλλεγούν έπιπλα, εξοπλισμό, τρόφιμα για τους πρόσφυγες που επανεγκαθίστανται. Όλες αυτές οι οργανώσεις και οι θρησκευτικέ και οι μη θρησκευτικέ υποστηρίζουν όλους τους πρόσφυγες ανεξάρτητα από τη θρησκεία των προσφύγων. Το Υπουργείο Υγείας επίσης χρησιμοποιεί μη κυβερνητικού φορείς όπως και το Υπουργείο Εξωτερικών για να παρασχεθούν υπηρεσίες αλλά το μεγαλύτερο μέρος των υγειονομικών υπηρεσιών δίδεται μέσω των πολιτιακών κυβερνήσεων και στη συνέχεια διανέμεται σε τοπικό επίπεδο, σε κυβερνητικού και μη κυβερνητικούς φορείς. Περιλαμβάνονται θέματα όπως εκπαίδευση για, για την αγορά εργασίας, εκπαίδευση στα αγγλικά και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν προγράμματα για πρόσφυγες με ειδικές ανάγκες. Μια τρίτη πτυχή που θα ήθελα να υπογραμμίσω και πάλι είναι κάτι το οποίο ανέφερε προηγουμένως ο είναι το θέμα της οικονομίας κλίμακος, των οικονομιών κλίμακος. Μιλήσαμε για τους αριθμούς που επανεγκαθίστανται στις ΗΠΑ. Το γεγονός ότι έχουμε μεγάλους αριθμούς, αυτό μας επιτρέπει να διοργανώσουμε το πρόγραμμά μας με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Έχουμε 8 κέντρα επανεγκατάσταση σε όλο τον κόσμο που μας βοηθούν στην επιλογή και τον έλεγχο των ε, προσφύγων αυτών. Και αυτό σε συνεργατικές συμφωνίες με ΜΚΟ που συνεργάζονται και κάποια από αυτά τα κέντρα είναι μεγάλα κέντρα. Κάποια από αυτά, όπως πρώτο, στην Ναϊρόμπι, έχουν πάνω από 200 εργαζόμενους και καλύπτουν ευρείες γεωγραφικές περιοχές. Με το να έχουμε αυτά τα περιφερειακά κέντρα, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το κόστος επεξεργασίας για τους πρόσφυγες. Μπορούμε να κρατήσουμε ένα μεγάλο αριθμό μελών του προσωπικού με τις κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες και να χρησιμοποιούμε και να μεταλαμπαδεύουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Ακόμα και αν δεν έχει κάνει τόσο μεγάλη κλίμακα, υπάρχει η δυνατότητα σε εθνικό επίπεδο να έχει κάνει οικονομία κλίμακος, με το παράδειγμα του χάρη να έχει ένα <clears throat> σταθερό πρόγραμμα ποσοστώσεων και όχι μονάχα ad hoc επανεγκατάσταση και το να υποστηρίζει μεγαλύτερες ποσοστώσεις που προωθούν την οικονομία ε, κλίμακος. Αυτά τα λέω μετά από την εμπειρία μου, έχοντα συζητήσει με άτομα που εμπλέκονται σε αυτέ τι διαδικασίε στι ΗΠΑ και στην Ευρώπη και πράγματι είναι πιο εύκολα από κάποιε άποψει να επαναγκαταστήσει κανεί μεγάλου αριθμού προσφύγων και όχι μικρότερου. Με το να έχει κανεί μια σταθερή ποσόστοση, αυτό επιτρέπει για να υπάρχει σχεδιασμό, να υπάρχουν επαφέ με όλου του εμπλεκομένου και να υπάρχει ένα σχεδιασμό για τη συνέχιση του προγράμματο στο μέλλον και μπορούν τα προβλήματα να εντοπιστούν σε ένα πρώιμο στάδιο. Όταν έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα με μεγάλους αριθμούς, αυτό επιτρέπει να διατηρηθεί επαφή με τις τοπικές κοινότητες, με τους ε, ιδιοκτήτες ε, καταλημάτων, με τους εργοδότες, ώστε δεν χρειάζεται κάθε φορά που έχετε κάποιος καινούριος να ξαναρχίσει κανείς από την αρχή. Και δημιουργείται και μια εμπειρία σε αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τον τομέα αυτό που μπορούν να αντιμετωπίσουν έτσι καλύτερα τα προβλήματα όταν ανακύπτουν. Κάτι ακόμα όμως το οποίο με εντυπωσίασε είναι ο βαθμός στον οποίο με το να έχουμε μεγαλύτερους αριθμούς επαναγκαθισταμένων μπορούμε να έχουμε μικροκοινότητος των ατόμων αυτών που μπορούν να δώσουν αλληλοβοήθεια ο ένας στον άλλο και μπορούν να βοηθήσουν αυτούς που έρχονται οι παλιότεροι εγκατεστημένοι να βοηθήσουν σε παιδική παραδείγματος χάρη φροντίδα ή σε δημιουργία θέσεων εργασίας και υπάρχει και ένας βασικώς μια δεξαμενή ατόμων που έχουν τις κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες για να βοηθήσουν τους νέο ερχόμενους σε αυτές τις περιοχές. Μπορούν λοιπόν οι επανεγκαταστηθέντες να βοηθήσουν και τους άλλους όταν παρίσταται η ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τόμας. Βεβαίως οι αριθμοί των ΗΠΑ όσον αφορά τη μεταγκατάσταση είναι εντυπωσιακοί, αλλά το ίδιο το πρόγραμμα είναι το πιο εντυπωσιακό ο τρόπος με τον οποίο καταφέρει να παντρεύει τα ωφέλη ε, και τα ε, το, το συμφέρον των κοινοτήτων. Ε, είχαμε μία πρώτη βίντεο διάσκεψη για την επανεγκατάσταση με την Ουάσιγκτον και πραγματικά είδαμε πώς γίνεται η δουλειά αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα περνάμε στον εκπρόσωπο της Δανίας, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα της μετεγκατάστασης και που θα μας δείξει πόσο σημαντικό είναι το θέμα της επανεγκατάστασης ε, για τις χώρες μέλη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίδεται αυτή η ευκαιρία να ασχοληθώ ε, με αυτό το θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Εγώ παρακολουθώ το θέμα της επανεγκατάστασης ε, από την ε, αρχή. Γνωρίζετε ότι η Δανία πρόσφατα απέκτησε νέα κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε κάποιες αλλαγές όσον αφορά ε, το θέμα της ε, μετεγκατάστασης ε, και έχει ήδη προαναγγείλει η κυβέρνηση ότι θα αλλάξει τα κριτήρια επιλογής όσον αφορά την μετεγκατάσταση και ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο μέλλον. Αυτή η αλλαγή γίνεται έτσι ώστε να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες ε, σε όλους. Ε, δεν θα αλλάξει όμως το, η ποσόστοση ε, των 700 ατόμων των 500 με 700 ατόμων κάθε χρόνο. Και επίσης χαιρόμαστε που το θέμα αυτό αποτελεί και μέρος της σημαντικής ακρόασης του Κοινοβουλίου. Το 1978 ξεκίνησε το δανέζικο σύστημα επανεγκατάστασης και βεβαίως διέπεται από διεθνεί συμφωνίες. Ε, οι πρόσφυγες αυτές αναφέρονται ως quota refugees, ε, δηλαδή σαν, ε, σαν πρόσφυγες της, της ποσόστοσης. Το ε, έγιναν κάποιες ε, τροποποιήσεις ε, του νομικού πλαισίου και φτάσαμε περίπου στα 500 άτομα το χρόνο και βεβαίως το, η ποσόστοση αυτή είναι ευέλικτη. και ε, επίσης έχουν συμπεριληφθεί πλέον μετά από την τροποποίηση και του 2005 ε, και ε, άτομα τα οποία πλέον επιλέγονται με νέα κριτήρια επιλογής τα οποία είναι εποφελία και της Δανίας και των ετούντων. Θέλω να πω δηλαδή ότι διευκολύνεται με τον τρόπο αυτό η ένταξη των ατόμων στην κοινωνία. Ε, και πλέον θα δίνεται μεγαλύτερη σημασία στην προστασία των προσφύγων. Ε, ο κύριος στόχος ε, είναι να υπάρξει δανέζικης πολιτικής επανεγκατάστασης ε, είναι βεβαίως να προστατεύονται οι πρόσφυγες. Επίσης, ε, στην ε, Δανία πλέον έχουμε επίγνωση όλο και περισσότερο τη στρατηγική σημασία που μπορεί να έχει η επανεγκατάσταση και η δυνατότητα παροχής επιλογών και δυνατοτήτων στους πρόσφυγες και βεβαίως ε, είναι δυνατή πλέον η διαπραγμάτευση της επανεγκατάστασης έναντι προσφοράς προς την, ή ανταλλαγμάτων προς την ε, κοινωνία. Από το 2005 ε, στην Δανία υπάρχει ένα σύστημα ε, προ-εγκατάστασης ε, και μετά μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεγκατάστασης ακολουθούν οι πρόσφυγες ένα πρόγραμμα ένταξης στην κοινωνία. Το σύστημα επανεγκατάστασης ε, στη Δανία αφορά τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Ε, αυτοί τα άτομα τα οποία επιλέγονται στις διαδικασίες επιλογής, ε, αυτά τα οποία εμείς ονομάζουμε expedited cases, δηλαδή τις πιο επίγουσες περιπτώσεις όταν υπάρχει κίνδυνος άμεσης επαναπρόθεσης, καθώς επίσης και μια τρίτη κατηγορία που αφορά ανθρώπους που χρήζουν άμεσης εφροντίδας, παροχή ιατρικής βοήθειας κτλ. Στη διάρκεια των ε, αποστολών, ε, μέλη της Δανέζικης Αντιπροσωπείας έρχονται σε επαφή και παίρνουν ε, συνεντεύξεις στα άτομα έτσι ώστε να επιλέξουν τις, περιπτώσεις υποθέσεις αυτές. Μετά γίνεται η παρουσίαση στην Υπηρεσία Μετανάστευσης. Η Υπηρεσία έρχεται σε επαφή με μη κυβερνητικές οργανώσεις και προχωράει η διαδικασία. Η υπηρεσία μετανάστευσης τελικά είναι υπεύθυνη για την τελική απόφαση και για γενικές αλλά και για ε, επιμέρους ε, περιπτώσεις. Ε, στις, στη δεύτερη περίπτωση, τις ε, επίγουσες δηλαδή υποθέσεις, στις οποίες η επαναπρόθεση είναι πολύ πιθανή, εκεί γίνεται μια επίγουσα διαδικασία έτσι ώστε να, να σταματήσει η διαδικασία επαναπρόθεσης. Η τρίτη κατηγορία, αυτή που ονομάζουμε εμείς 20 και πλέον, 20 or more, αφορά 20 με 30 άτομα κάθε χρόνο. Ε, και βασίζεται σε φακέλους τους, έχει, οποίους έχει υποβάλει η ύπατη αρμοστία ή που έχουν επιλέξει σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία ή οι αποστολές ε, το, τη της ε, Δανίας. Όσον αφορά τώρα τα κριτήρια ε, επιλογής, πρώτον θα πρέπει το άτομο να θεωρείται πρόσφυγα σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία. Επίσης θα πρέπει να καλύπτει τα κριτήρια διεθνούς προστασίας ή ανθρωπιστική ανθρωπιστικού στάτους υπό τον δανέζικο νόμο σε αυτή την περίπτωση ε, η υπηρεσία μετανάστευσης της Δανίας ε, θα ελέγξει το κατά πόσον ε, τα άτομα αυτά μπορούν να λάβουν τελικά μια κάρτα παραμονής, αλλά αυτό ενδεχομένως τώρα και να αλλάξει. Επίσης υπάρχει και η κατηγορία η οποία ελέγχεται σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες, συνθήκες υγείας κτλ. Ε, στην ε, ε, κατηγορία των ατόμων που η υπόθεσή τους εξετάζεται έτσι ώστε να τους δοθεί ενδεχομένως άδεια παραμονής. Λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική κατάσταση, το, ο βαθμός ε, μόρφωσης και τα λοιπά. Πριν, από την, πριν ληφθεί η τελική ε, απόφαση θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, υποβληθεί ο ενδιαφερόμενος σε ιατρικές εξετάσεις. Τρει, τρεις αποστολές αναέτος γίνονται αποστολές επιλογής. Πάντα από το Υπουργείο γίνεται η... Από Υπουργείο γίνεται αυτό προτάσει της υπηρεσία μετανάστευση. Αυτή η σύσταση βασίζεται σε διμερείς ε, επαφές και επίσης σε διαβουλεύσεις οι οποίες γίνονται σε ευρύτερο επίπεδο μέσα σε μια ομάδα εργασία. Η ομάδα εργασίας για τα θέματα αυτά έχει ε, συνεργασία με την ύπατη αρμοστία για, την, για τους πρόσφυγες και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε μια πολιετή δέσμευση για να προστατεύσουμε τους ε, πρόσφυγες και να αυξήσουμε τη δυνατότητα επανεγκατάστασης. Το 2008 ε, αντιμετωπίσαμε χώρες όπως η Μαλαισία, Ζάμπια και Νεπάλ. 2009 το Νεπάλ και η Μαλαισία αλλά και η Ρουάντα για να αντιμετωπίσουμε πρόσφυγες από το Κονγκό το Νεπάλ για τους ε, πρόσφυγες από το Βουτάν και η Μαλαισία για τους, ε, επίσης για τους ε, πρόσφυγες από την Βερμανία. Στη συνέχεια είχαμε αποστολές επιλογής στο Νεπάλ και στην Κένια. Αυτό ήταν 2010 και το 2011 έχουμε, κάναμε επιλογές στο Νεπάλ, στη Ζιμπάμπουε και στη Μαλαισία για τους πρόσφυγες από το Μπουτάν, από τη Βερμανία και τη Δημοκρατική Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτά λοιπόν για το 2011. Για το 2012 θα αποφασίσουμε αργότερα ή στις αρχές του 2012. Εν τέλει, οι μελλοντικέ προοπτικές. Βλέπουμε ότι στρατηγικά μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο η επανεγκατάσταση στην πολιτική ασύλου και μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει ρεαλιστικά αντιμετώπιση των προσφυγικών ρευμάτων, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία στην εγγύης περιοχή από που, σε εγγύης περιοχές από όπου προέρχονται οι πρόσφυγες. Πρέπει να αυξηθεί λοιπόν με αυτή την χρήση η παγκόσμια δυνατότητα προστασίας. Είναι ένα εργαλείο λοιπόν το οποίο θα βοηθήσει την παγκόσμια δυνατότητα προστασίας και αυτό κάνουμε εδώ και μία δεκαετία προσπαθώντας να προχωρήσουμε προ την κατεύθυνση αυτή. Εμεί υποστηρίζουμε τα περιφερειακά προγράμματα προστασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίζουμε λοιπόν σημαντικό ρόλο στο να προωθήσουμε τέτοιε τοπικέ πρωτοβουλίε, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορούν με την επανεγκατάσταση να βοηθήσουν τι χώρε να ενισχύσουν την ικανότητά του για να προστατεύσουν του πρόσφυγες και με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις βασικές αιτίες των προβλημάτων, να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ε, επίγνωση και να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των πολιτών τους. Η δημιουργία ικανοτήτων έχει τεράστιο διδακτικό και παιδαγωγικό αποτέλεσμα που μπορεί να βοηθήσει τις χώρες αυτές και μπορεί να είναι συμπληρωματική άλλων μορφών ανάπτυξης. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και να ενισχύσουμε την γενική ικανότητα προστασία ατόμων που χρειάζονται διεθνή προστασία. Μπορούμε λοιπόν με τον τρόπο αυτό να έχουμε μεγαλύτερη ικανότητα των περιφερειών και υψηλότερα πρότυπα για να είναι πιο αποτελεσματική η αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Πιστεύω ότι αυτή η ιδανική εμπειρία μπορεί να σας φανεί χρήσιμη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλίνστρουπ. και είναι πάρα πολύ θετικά αυτά που λέτε. Η ιδανική αυτή εμπειρία μπορεί να παίξει πραγματικά παιδαγωγικό και διδακτικό ρόλο και για μας και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό η ιδανική προεδρία να μπορέσει να αυξήσει την συνειδητοποίηση όλων στο Συμβούλιο και να μεταλαμβατεύσει αυτό το μήνυμα το οποίο μας παρουσιαστεί εδώ Έχουμε δει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ένα από τα πιο σημαντικά εγχειρήματα είναι το να αυξάνεται η συνειδητοποίηση όλων για να μπορέσει να προωθηθεί η συζήτηση αυτή για την επανεγκατάσταση. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για αυτά που μας είπατε για τη δανεική εμπειρία. Δεν θα κάνω σχόλια καταληκτικά, γιατί έχω ήδη κάνει σχόλια. Απλώς θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στη συζήτηση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Τα καλά νέα είναι ότι έχει εγκριθεί το σχέδιο αυτό για την ε, επανεγκατάσταση, το έκτακτο σχέδιο επανεγκατάστασης και το σχέδιο αυτό για τους Δήμους. Έχουμε λοιπόν μια μεγαλύτερη επίγνωση και συνειδητοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Και όπως είπε και η Κομισιόν, μπορούμε το 2012 να εντείνουμε αυτές τις προσπάθειες. Και πρωτού ξεκινήσουμε την ε, ανταλλαγή απόψεων, θέλω να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για την υποστήριξή της, υποστήριξή της για τα θέματα αυτά. Ο Αντώνιο μας ο πρώτος ο οποίος ζητάει το λόγο πολύ σύντομα γιατί έχουμε φτάσει και στα συμπεράσματα άλλωστε. Ήθελα να ευχαριστήσω για την ηθική δίδαχη που μας έγινε σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά σε πρακτικό επίπεδο, όπως είπε πολύ καλά και ο πρόεδρος ε, Ταβάρες, θα ήθελα από εδώ να σταλεί και πάλι το μήνυμα ότι το κέντρο της Ευρώπης, ε, οι Βρυξέλλες, η πρωτεύουσα της Ευρώπης, τα θεσμικά μας όργανα αποστέλουν το μήνυμα του κατεπήγοντας που είπε ο πρώτος ομιλητής για τους 5.000 πρόσφυγες στη Βόρεια Αφρική που πρέπει απευθείας το συντομότερο δυνατόν να λάβουν την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτοί οι 5.000 θα ήθελα να διευκρινίσω το εξή. Είναι ήδη 4.000 περίπου 5.000 πρόσφυγες που έχουν ταξινομηθεί στο παλιό γραφείο της Τρίπολης και έχουν βρεθεί ε, κάποιοι στη Λαμπεντίουσα, κάποιοι στη Σούσα. Είναι αυτοί οι 5.000 ή υπάρχουν άλλοι 5.000 διαφορετικοί τους οποίους θα προσθέσουμε σε αυτούς τους οποίους ήδη έχουμε στον κατάλογο και θα πρέπει να υποδεχθούμε ως πρόσφυγες ε, και έχουμε και την ηθική υποχρέωση ως Ευρωπαϊκή Ένωση να τους ε, υποτεχθούμε. Έχουμε άλλους 5.000 που προστίθενται στο πρόβλημα της ε, Σούσα ή ε, είναι οι ίδιοι. 10.000 ή 5.000. Η Τζιν Λάμπερ τώρα. Ευχαριστώ. Ένα από τα θέματα τα οποία προέκυψαν συνεχώς όταν συζητούσαμε τα θέματα πολιτικής ασύλου με κάποια κράτη-μέλη είναι οι ανησυχίες που υπάρχουν ε, σε θέματα επανένωσης οικογενειών. Ότι αυτή τη στιγμή ανοίξει πόρτα για τους ένα-δύο πρώτους, από εκεί και πέρα έρχονται όλοι. Όσον αφορά την επανεγκατάσταση λοιπόν, προκύπτει το θέμα της επανένωσης. Μας ανησυχεί και αν ναι, Πώς αντιμετωπίζετε. Ξέρω τι λένε οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτού και ξέρω ότι πολλά κράτη-μέλη δεν ε, το τηρούν όπως πρέπει. Αλλά θα ήθελα να ακούσω τι επιχειρήματα χρησιμοποιούνται για το θέμα αυτό. Δεν ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Δεν ξέρω αν κάποιο ε, θέλει να απαντήσει τα δύο ερωτήματα που ετέθησαν. Όσον αφορά τους 5.000, ο κύριος Έτια Μεζιάν, κάποιοι από αυτούς τους ετούντες άσελο Κάποιοι ε, αποτέλεσαν αντικείμενο του γραφείου της Λιβύης, αλλά ε, Κατόπιν έκλεισε αυτό το γραφείο και υπήρξαν ακόμα και πρόσφυγες από τον Ταρφούρ στη Λιβύη που δεν ε, είχαν πρόσβαση στο γραφείο στη Λιβύη λόγω της κατάστασης της ΥΠΑ της Αρμοστίας στη Λιβύη. Πρόκειται λοιπόν ένα ε, μείγμα ανθρώπων. Κάποιοι είχαν αναγνωριστεί, κάποιοι δεν είχαν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες, κάποιοι μπόρεσαν να φτάσουν στα γραφεία μας στη Λιβύη και αυτή τη στιγμή πέρασαν τα σύνορα και έφτασαν στο στρατόπεδο της Σούσα, ε, τους εξετάσαμε αναπερίπτωση. Κάποιοι αναγνωρίζονται και ε, αντιμετωπίζονται λίγο διαφορετικά από αυτούς που δεν έφτασαν ποτέ στο γραφείο μας. Για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα λοιπόν. Υπάρχει αυτή η ομάδα των 4 με 5.000 ανθρώπων που αυτή τη στιγμή είναι ε, κάποιοι αναγνωρισμένοι και κάποιοι άλλοι όχι. Υπάρχει και μια ε, ομάδα ανθρώπων στη Λιβύη και ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες σύντομα στη Λιβύη του γραφείου μας και ελπίζω ε, ε, να μπορέσουμε να ασχοληθούμε και με αυτούς που βρίσκονται στη Λιβύη. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αναφερόμαστε σε πρόσφυγες που φτάνουν μαζί με μετανάστες στη Λαμπεντούζα, όπως μας είπατε. Ορισμένες φορές ε, διστάζουμε να πούμε ότι ξεκινήστε με την επανεγκατάσταση γιατί επηρεάζει την κανονική ροή ανθρώπων. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο διαφορετικές ομάδες. Ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα στρατόπεδα προσφύγων και κάποιοι άλλοι που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για ανθρώπους που επέστρεψαν από την Τινησία στη Λιβύη για να πάρουν τα διαβατήριά τους και με να πάρουν στη συνέχεια σκάφη λαθρεμπόρων για να πάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Λαμπεντούζα, ε, γιατί δεν μπορούσαν να περιμένουν την επανεγκατάσταση. Μετά από την κατάσταση το Μάιο, τη φωτιά, ένιωσαν ότι δεν είναι ασφαλής και θέλησαν να πάρουν ένα καράβι και να φύγουν. Ε, ε υπάρχει λοιπόν το θέμα της μεγάλης διάρκειας της επανεγκατάστασης και ε, υπάρχει περίπτωση να επιλέξουν λοιπόν οι πρόσφυγες να ακολουθήσουν τις πορείες των δουλεμπόρων. Όσον αφορά τώρα την ερώτηση της κυρίας Λάμπερτ, Νομίζω ότι και η κυβέρνηση της Δανίας θα πρέπει να απαντήσει κατά πόσον τους δημιούργησε πρόβλημα το θέμα της επανένωσης των οικογενειών μετά από την επανεγκατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα για να ε, βρούμε την ταυτότητα των ανθρώπων που ε, πρέπει να επανεγκατασταθούν και θέλουμε να επανανήσουμε την οικογένεια. Γι' αυτό λοιπόν φροντίζουμε οι πρόσφυγες που παρουσιάζονται ε, ως οικογένεια είναι πράγματι οικογένεια. Αν λένε ότι ε, πει για παράδειγμα μια γυναίκα σε κίνδυνο ότι ο άντρας της εξαφανίστηκε, ε, φροντίζουμε ε, να βεβαιωθούμε ότι ο σύζυγός της δεν μένει στην άλλη πλευρά του στρατοπέδου για παράδειγμα. Ε, στα τόσα χρόνια που έχουμε επανεγκατάσταση υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και αίτημα επανένωσης με τη αμέλη της οικογένειας αργότερα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει δημιουργήσει προβλήματα στην επανεγκατάσταση αυτή καθ' αυτή. Πολύ σημαντικό, ο κύριος Σταβάρες, για τα θέματα της επανεγκατάστασης είναι ε, πώς μπορούμε να απομακρύνουμε ανθρώπους από τους δουλεμπόρους ε, και το πώ μπορεί να είναι ζήτημα ζωής και θανάτου το γεγονός ότι δεν αναπτύσσονται καταλήλω οι πολιτικές. Και αυτό το είδαμε ε, στη Μεσόγειο πρόσφατα. Και το ερώτημα τη κυρία Λάμπερτ. Παρουσιάστηκε η εμπειρία της υπάρχει αρμοστίας με τους πρόσφυγες που έχουν μια μεγαλύτερη εμπειρία για την αντιμετώπιση αυτή, αλλά και εμείς σαν χριστιανικός φορέας ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για τα θέματα της οικογένειας και το πόσο καλά είναι τα πράγματα ή δεν είναι εξαρτάται από το αν ρωτάτε τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ή τις κυβερνητικές αρχές. Για μένα το πρώτο είναι το εξή όταν υπάρχει διαβεβαίωση, όταν υπάρχει η βεβαιότητα για την ε, σύνθεση της οικογένειας, έρχονται πολλές φορές οι πρόσφυγες με πάρα πολλές ε, πολλά μηνύματα που του έχουν δώσει. Μην πείτε ότι έχετε οικογένεια, πείτε ότι έχετε μικρή οικογένεια στην αρχή θα σα αφήσουν να πάρτι μονάχα λίγα άτομα. Αυτό κάνει πολύ δύσκολη την κατάσταση στην αρχή. Όσο καλή και να είναι η υπεύθυνη τη της τη αρμοστία για να καταλάβουν ποιο ανήκει και ποιο ανήκει σε μια οικογένεια. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, ιδίω σε μια κατάσταση ενό μεγάλου καταβλισμού σε συνθήκε έκτακτε. Δεν έχετε το χρόνο να το κάνετε αυτό. Και στη συνέχεια βλέπουν οι επιτόπιοι φορείς ότι <clears throat> υπάρχει και ένα άλλο παιδί, υπάρχει κάποιο άλλο μέλος οικογένειας το οποίο δεν το έχουν αναφέρει ακριβώς γιατί ο πρόσφυγα λέει ότι μου είπαν ότι πρέπει να είναι μικρή οικογένεια δεν θα με πάρουν. Και στη συνέχεια τι ακριβώς περιλαμβάνει η οικογένεια. Αυτό είναι ένα θέμα στην Κένια υπήρχαν πολλά ορφανά τα οποία στη συνέχεια τα υιοθετήσανε οι οικογένειε, αλλά δεν ήταν ε, με την κλασική έννοια. Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι αυτή δεν είναι η οικογένειά του, αλλά στην πράξη τα παιδιά αυτά ζουν με τους ε, ανθρώπους αυτούς για δεκαετία, για δέκα χρόνια χάρη. Όταν μπει λοιπόν κανείς στα θέματα της ε, οικογενικής επανένωσης, θέλετε το θέμα του νομικού ε, του νομικού καθεστώτος, αλλά ξέρουμε ότι σε πάρα πολλές χώρες ότι οι πρόσφυγες ίσα ίσα τα βγάζουν πέρα και είναι πολύ δύσκολο για αυτούς για να φέρουν κάποιο άτομο παραπάνω. Και είναι σημαντικό να υπάρξει κάποια δυνατότητα να έχουν οι άνθρωποι αυτοί την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν την οικογενειακή τους επανένωση. Αλλά παραμένει όλο αυτό ένα τεράστιο και δύσκολο θέμα. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα αυτό το θέμα της οικογένειας. Εμείς πάντα τους πληροφορούμε για το θέμα της οικογενειακής επανένωσης, ώστε να ξέρουν τι μπορούν να περιμένουν όταν έρθουν στην Δανία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχετε διαφορετικές έννοιες του τι αποτελεί μια οικογένεια. Είναι χρήσιμο και απαραίτητο να τους πληροφορούμε επακριβώς για να ξέρουν τι ακριβώς προβλέπεται. Και εμείς δεν διαχωρίζουμε τις οικογένειες. Όταν κάνουμε αποστολές επιλογής. Μπορεί να έχουμε τα παιδιά και τους, τα μωρά και τους ε, υπερήλικες να έχονται στην ίδια οικογένεια στη Δανία. Και όπως είπε και ο Τόρστεν, έχουμε πολλές φορές παιδιά που ζουν με γονείς μέσα σε εισαγωγικά, ανθρώπους που δεν είναι οι γονείς τους, αλλά απλώς τα έχουν υιοθετήσει. Και το δεχόμαστε και αυτό. Τους βλέπουμε σαν μια οικογένεια, σαν ένα οικογενειακό σύνορο. είναι, μπορεί να είναι μια οικογένεια η οποία έχει συστηθεί για αυτόν μονάχα το στόχο της ε, επιλογής. Αλλά όταν τα παιδιά ζουν με ανθρώπους για πολύ καιρό θα πρέπει να τους θεωρήσετε μια οικογένεια. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω κύριε Τόμας αν θέλει να προσθέσει κάτι. Όχι. Εντάξει. Αν δεν θέλει κανείς το λόγο. Έχουμε τελειώσει πριν από την ώρα μας. Και θα έχουμε περισσότερο χρόνο για τα συμπεράσματα και σε αυτό το κομμάτι θα προεδρεύσει η κυρία Τζιν Λάμπερτ. Ευχαριστώ Τζιν. Okay. Um, Ωραία. Ξέρω ότι για πολλούς λόγους ε, είναι αργά, οι περισσότεροι θέλουν ε, να φύγουν, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ένα επίσημο κλείσιμο κατά κάποιο τρόπο της ε, ημέρας. Βεβαίως ε, όλη αυτή η σημερινή ημέρα ήταν εξαιρετικά ε, αξιόλογη με πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις, πολλές πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν, μας βοήθησαν ήδη δηλαδή να δούμε με οριζόντιο τρόπο τη διασύνδεση πολλών θεμάτων. και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε οριζοντίως να μελετήσουμε κάποιες προτάσεις. Θα ζητήσω βεβαίως τώρα από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να πούν αν θέλουν δύο λόγια για να μας πούν την άποψή τους. Ε, θα έχω και εγώ δύο λόγια να πω εξ ονόματος του Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν θέλει να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε σήμερα. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εκδήλωση. Ακούσαμε πολλά, παρακολούθησα, παρακολουθήσαμε ε, όλα τα σχόλια, ακόμα και τα επικριτικά σχόλια και τα αρνητικά κατά κάποιο τρόπο σχόλια. Ε, είναι πραγματικά ενδιαφέροντα και πάνω σε αυτά θα δουλέψουμε τους επόμενους μήνες, εβδομάδες και μήνες. κατά τα λοιπά. Στρεφόμαστε προς το μέλλον, λέτε. Ε, ο στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δεύτερη γενιά νομοθεσία είναι να βελτιωθεί ο συντονισμός και η συνοχή ανάμεσα ε, στα διάφορα ε, στις διάφορες γενιές και στα διάφορα νομοθετικά έγγραφα. Επίσης θα θέλαμε ε, να, με τις ε, νέες μας ε, προτάσεις θα θέλαμε να ενυψώσουμε λίγο το επίπεδο των προτάσεων και να βελτιώσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία. Βεβαίως εμείς ακολουθούμε μία προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και πλέον βρισκόμαστε και στην αντίληψη των κοινών ε, στάνταρ. Κατανοούμε βεβαίως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλήσεις και διαφορές ε, και επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στρέφεται ε, εν προκειμένου προς τους δύο συνομοθέτες, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας την στήριξή τους έτσι ώστε να επιτευχθούν αυτά τα υψηλά πρότυπα. Η Πολωνική Προεδρία ήταν πραγματικά πάρα πολύ δραστήρια και η Κομισιόν θέλει να την ευχαριστήσει γι' αυτό. Και προσδοκούμε ότι θα έχουμε καλή συνέχεια των μελλοντικών εργασιών. Βεβαίως φαντάζομαι ότι όλοι κατανοούν ότι χρειάζονται και θα χρειαστούν ε, οπωσδήποτε ε, κάποιοι συμβιβασμοί έτσι ώστε να καλύψουμε ε, και την, ε, το χρονικό περιθώριο του 2000, τη χρονική προθεσμία του 2012. Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι όλοι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε κάτι και ε, επομένως ε, άποψή μας είναι ότι το πλαίσιο θα πρέπει να έχει ε, σαφές πλαίσιο, καθαρό, κατανοητό πλαίσιο, έστω και αν κάποια προβλήματα μπορούν να διορθωθούν. Αυτά νομίζω, δεν υπάρχει λόγος να πω τίποτα άλλο. Να τελειώσω λέγοντας ότι φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι στη διάθεση των δύο συνομοθετών, Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, από την άλλη πλευρά βασιζόμαστε σε σας, περιμένουμε από σας. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσω στο συνομοθέτη μου τελικώς, ε, ο κύριος Σώστακ. Θα μιλήσει από πλευράς ε, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων ε, του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Ε, δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Δεν έχουμε χρόνο να διατρέξω και τα επτά τμήματα της συνεδρίασης να σταθώ καταρχάς στην εξωτερική διάσταση της πολιτικής, επανεκα... της ε, πολιτικής ασύλου. Κάναμε ενδιαφέρουσα συζήτηση για την επανεγκατάσταση και όλοι αναγνωρίζουν ότι η επανεγκατάσταση είναι μία από τις πολύ σημαντικές πτυχές ε, της ε, πολιτικής ασύλου. Είναι ένας από τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται τα κράτη-μέλη επιθελουσίας βάσεως, Λίγα κράτη-μέλη έχουν προγράμματα κατάστασης αυτή τη στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αδρανής. Ε, υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης ε, και ε, βάσει του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και ελπίζουμε να επεκταθούν αυτές οι δυνατότητες στις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές. Όπως υπόθηκε υπάρχει μια πρωτοβουλία επιτάπητος αυτή τη στιγμή, αλλά δυστυχώς υπάρχουν διαφωνίες ε, για τις εφαρμοστές διαδικασίες και καθυστερούει και λόγω των ε, διοργανικών ε, σχέσεων και δεν έχει υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αλλά μας ενδιαφέρει η εξέβρεση συμβιβασμού. Και να σας πω ότι υπάρχει δέσμευση από πλευράς πολιτικής Προεδρίας για να προχωρήσουν τα θέματα αυτά. Η δεύτερη μου παρατήρηση αφορά τις ε, εσωτερικές πτυχές της πολιτικής ασύλου και νομίζω ότι είναι πιο ουσιώδης λόγω και της σημερινής ακρόασης. Τα μέλη του Συμβουλίου και βεβαίω η Προεδρία συμφωνούν ότι το σύστημα ασύλου των κρατών μελών πόρο απέχουν από την τελειότητα. υπάρχουν μέλη του Συμβουλίου και η Προεδρία που συμφωνούν ότι κάποια κράτη-μέλη χρειάζονται και την αρρωγή μας. Γι' αυτό ακριβώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, τα 27 κράτη-μέλη, ε, με συνένεση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει ανάγκη για ένα κοινό σύστημα σύλλου μέχρι το τέλος του 2012. Αυτό επαναεπιβεβαιώθηκε τον Ιούνιο άλλωστε. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι είναι παντού χαμηλές προδιαγραφές στα κράτη-μέλη. Κάθε άλλο. Ακούσαμε κάποια παραδείγματα για τις χειρότερες δυνατές πρακτικές, για τις γλώσσες, για τα πρότυπα και τη διερμηνία, αλλά ακούσαμε πολύ λιγότερα για τις καλύτερες πρακτικές στον τομέα αυτό, οι οποίες υπάρχουν. Ακούσαμε ένα παράδειγμα ε, για ένα νησί στο οποίο... Ε, οι εγκληματίες ε, μπαίνουν ε, δίπλα στις γυναίκες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ε, υπάρχουν μόνο αυτά τα παραδείγματα. Υπάρχει οδηγία η οποία προβλέπει να μην υπάρχει αντίστοιχο φαινόμενο και υπάρχει και δυνατότητα ελέγχου στους χώρους κράτησης ώστε να ελέγχουν ότι τηρούνται οι κανόνες. Υπάρχει και το παράδειγμα που ακούσαμε κάποιου που συμπεριφέρεται σαν αστυνομικός και μάλιστα με υποχθόνιες σκοπούς και κάποιοι εργάζονται με πολύ μεγάλη πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με πολύ μικρό προϋπολογισμό. Γιατί σας τα λέω αυτά. Γιατί ε, αφορούν τις διαπραγματεύσεις για τα θέματα του ασύλου και ιδίως την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου. Οι διαπραγματεύσεις για την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Καταρχάς, Έχουμε 27 πολύ διαφορετικά συστήματα σύλλου που δεν αναρμονίστηκαν ποτέ. Αυτή είναι η πρώτη απόπειρα εναρμόνισης. Κατά δεύτερον, η πρώτη γενεά ε, μέτρων ε, στον τομέα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε κάποια ελάχιστα πρότυπα, αλλά στην πράξη έχουν τεθεί σε εφαρμογή μόλις πριν από 1,5 χρόνο και ακόμα δεν είναι βέβαιο πώς ακριβώς ε, λειτουργούν. Τρίτον, ε, στην ε, περίπτωση της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου, πολλά από τα θέματα ε, πολύ συχνά αφορούν βασικές γενικές αρχές του αστικού δικαίου και των διοικητικών διαδικασιών των κρατών μελών και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αλλάξουμε. Επιπλέον, κάτι το οποίο νομίζω ότι ήταν πολύ σαφέ από τη συζήτηση για την κράτηση, πρόκειται για ένα τομέα τη νομοθεσία που ακόμα και βάσει τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ε, επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα. Για παράδειγμα, τη σύσταση του Συμβουλίου Υπουργών του Συμβουλίου τη Ευρώπη για την κράτηση. Δείτε το δεύτερο λόγο που αναφέρεται για την ανάγκη να υπάρχουν αποδείξεις ε, σε ένα φάκελο και πέστε μου κατά πόσον είναι απλή αυτή η διάταξη ε, αυτό που προσπαθούμε να κατανοήσουμε στη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων ε, γίνεται με πολύ μικρή βοήθεια από τα δικαστήρια ή από οποιονδήποτε άλλον. Τέλος, πολλά από τα πρότυπα που αναφέρονται στο κείμενο αυτό υπερβαίνουν τις εγγυήσει που έχουμε στη διάθεσή μας ε, για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους ίδιους και θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον είναι αιτιολογημένο να υπερβούμε τις εγγύησεις που δίνονται στους πολίτες των κρατών μελών ε, ε, προς όφελος ε, υπηκών τρίτων χωρών σε αυτές τις διαδικασίες ασύλου. Αν προσθέσουμε δε και τον πολύ στενό προϋπολογισμό, έχουμε μία πολύ πολύ περίπλοκη διαπραγμάτευση. Με άλλα λόγια, θεωρούμε ότι Εύκολα μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει τις διαπραγματεύσεις ε, ως έναν αγώνα προς τον πάτο και το γεγονός ότι το Συμβούλιο προσπαθεί να ρίξει ε, το επίπεδο και κάποιο άλλο θεσμικό όργανο προσπαθεί να ανεβάσει τα επίπεδα. Δεν ισχύει. Έχουμε ένα αμάλγαμα τελείως διαφορετικών καταστάσεων ασύλου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποια συστήματα ασύλου είναι πολύ καλά και υπάρχουν και πάρα πολύ δύσκολα νομικά μέσα και με όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να καταλήξει σε συμφωνία για το κείμενο αυτό μέχρι το τέλος του 2012, δηλαδή μέχρι το τέλος της συγκεκριμένη τριάδας προεδρών. Η Πολεωνική Προεδρία ε, όπως ακούσαμε και ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια, κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να δημιουργήσει την κατάλληλη όθηση για να προχωρήσουν τα θέματα αυτά. Συνεργαζόμαστε στενά με την επόμενη Δανική Προεδρία και με την ε, Κυπριακή Προεδρία. Και φυσικά, όπως είπαν όλοι, θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα στο τέλος. Η τελευταία μου παρατήρηση είναι, είναι ότι η Προεδρία είναι ισχυρή αν είναι ισχυρά και τα κράτη-μέλη που εκπροσωπεί. Αν θεωρείτε λοιπόν ότι η Πολωνική Προεδρία δημιουργεί μια θετική δυναμική, αυτό ισχύει και γιατί συνεργάζεται αγαστά με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε των δυσκολιών που υπάρχουν σε ορισμένα από τα θέματα αυτά. Και το Κοινοβούλιο φυσικά γνωρίζει και από το παρελθόν, από το, την εποχή που δεν ήμασταν νομοθέτες για τα θέματα αυτά, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν δυσκολίες στο Συμβούλιο. Πρέπει να πούμε κιόλας ότι ορισμένες φορές νιώθουμε ότι κάποιες από τις απαντήσεις που μας έχει δώσει το Συμβούλιο σε ορισμένα ερωτήματα, δεν θα πω σε ποιο Συμβούλιο ή ποιους εκπροσώπους του Συμβουλίου, νομίζουμε ότι συζητάνε για κάτι άλλο. Ότι αυτό είναι στοιχείο της δυσκολίας. Ότι πρέπει μερικές φορές να πείσετε κάποιους ότι υπάρχει ένα θέμα και μήπως πρέπει να συζητήσουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. για να εξασφαλίσουμε αυτή την προστασία που θα πρέπει να δίνει η νομοθεσία για τους. Δεν έχουμε πάντως καθόλου ψευδεστήσεις για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάθε κράτη-μέλη και για το πολιτικό κλίμα στο οποίο βρίσκονται και αυτοί από μας που έχουν ενδιαφέρον για τα θέματα του ασύλου θέλουν, θέλουμε πάντα να υπογραμμίσουμε την ανάγκη της προστασίας γιατί υπάρχουν κάποιες πολιτικές δυνάμεις Οι περισσότερες από αυτές ευτυχώς όχι σε θέσεις κυβερνητικές που θεωρούν ότι η παροχή ασύλου είναι ένα προνόμιο και όχι ένα ουσιαστικό δικαίωμα που αφορά τόσους πολλούς ανθρώπους. Θέλουμε λοιπόν όλοι να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε σχέση με το μέλλον που μπορούμε να προσφέρουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους στον πλανήτη που αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλα προβλήματα και που κινδυνεύουν να κινδυνεύουν από καταδίωξη ή από άλλες δυνατότητες να πληγούν. Θεωρούμε λοιπόν ότι <clears throat> αυτή η ακρόαση έχει βοηθήσει την προσπάθειά μας να λύσουμε κάποια από τα οριζόμενα, οριζόντια θέματα, για θέματα για ευάλωτα άτομα, για συνθήκες κράτησης κτλ. και θα θέλαμε μέχρι το 2012 να συμπληρωθεί η επεξεργασία των θεμάτων αυτών που συνάπτονται με το άσυλο. Δεν περιμένουμε θα γίνει αυτό τον Ιανουάριο του 2012, αλλά θα θέλαμε σίγουρα να γίνει το ταχύτερο δυνατό και να κλείσουν όλα αυτά τα θέματα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και κάποια από τα θέματα που <clears throat> δημιουργούν ανησυχία στα κράτη-μέλη για να επιτευχθεί η επέκταση των βελτίστων πρακτικών όπως αυτά που είδαμε πραγματικά για το Βέλιο σήμερα. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να επεκταθούν αυτές οι βέλτιστες πρακτικές από τα καλυτερα κάτι κράτη-μέλη στον τομέα αυτό. Και το άλλο το οποίο θέλω να πω, ξέρω ότι είσαστε επί ξηρού ακμής, αλλά έχουμε μία ψηφοφορία την επόμενη εβδομάδα για τα θέματα αυτά, για τα θέματα αναγνώρισης και αυτό είναι πραγματικά μια καλή είδηση. Θα, ας ελπίσουμε ότι θα εγκριθεί αυτό είτε με τους πίνακες αντιστοίχησης είτε όχι και όλα αυτά θα είναι μια σημαντική πρόοδος στο θέμα αυτό. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι συμμετέσχαν σήμερα στην ακρόαση, αυτούς που έμειναν όλη μέρα, αυτούς που συνέβαλαν στα διάφορα πάνελς και μας έδωσαν πληροφορίες, τους διερμηνείς και τους άλλους συνεργάτες που μας βοήθησαν. Ελπίζουμε όλοι λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα θέματα αυτά στην Ολομέλεια και ότι θα μπορέσει να δοθεί και μία ε, συνέχεια στην έκκλησή σας για τους 5.000 που θέλουν επαναγκατάσταση. Ευχαριστώ.